Okay, good morning, friends. We're about to start, but I'm going to invite Mr. Humble up to the... Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Να καλέσω τον κύριο Χάμπλ εδώ πάνω στο Προεδρείο. So, good morning, everybody. Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε. Αντίθετα με αυτά που ανακοινώθηκαν, εγώ θα προεδρεύσω τις ε, αυτή αυτής ε, και όχι ο Κλοντ ο οποίος ε, δυστυχώ δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να με ανεχτείτε σήμερα το πρωί. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που σήμερα θα συμμετέχουν 29 μέλη εθνικών κοινοβουλίων που εκπροσωπούν 14 κράτη-μέλη, περίπου τα μισά. Σίγουρα θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση και είμαι βέβαιη ότι του χρόνου θα συμμετέχουν όλα τα κρατημέλη. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Το σημερινό λοιπόν θέμα είναι η δημοκρατία και κρατός δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά αρκετά συχνά, γιατί η ευρωπαϊκή ενοποίηση και συνεργασία συχνά ορίζεται μέσω υλικών αγαθών και επιτευγμάτων. Αστυνομική συνεργασία, ενιαία αγορά. Συχνά λοιπόν ορίζεται μέσω οικονομικών όρων, αλλά συχνά ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση αξιών. Και αυτέ οι αξίε ουσιαστικά κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 των συνθήκων. Το οποίο είναι και το πιο σημαντικό στο άρθρο. Ενδεχομένω να θεωρήσει κανεί ότι το πιο σημαντικό είναι το άρθρο 1, αλλά Ουσιαστικά το πρώτο άρθρο αποτελεί ένα χαιρετισμό, στο δεύτερο άρθρο κατοχυρώνονται οι αξίε. Μα αυτέ οι αξίε λοιπόν έχουν αντιτυπωθεί με εξαιρετικό τρόπο. Είναι όμω ε, λόγια. Λόγια που έχουν γράψει οι διπλωμάτε, οι αξιωματούχοι, έχουν κάνει καλή δουλειά, δεν λέω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε την αίσθηση όλο και πιο πολύ ότι τα λόγια αυτά, το άρθρο αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη και θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνει όταν μιλάμε για κοινέ αξίε, τι σημαίνει. Έγινε ένα πρωινό εργασία πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζουμε τους νέους τρόπους μετανάστευσης, όπου και αναφέρουμε ότι νεοαφιχθέντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασπαστούν τις κοινέ μας αξίες. Ποιες είναι όμως αυτές οι κοινέ μας αξίες και ο ορισμός των κοινών αξιών αυτών δεν είναι απλή συζήτηση, ούτε είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα χρονικό διάστημα. Θα πρέπει διαρκώς να διεξαγάγεται σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα όλο και πιο πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό αποτελεί και τη βάση της συνεργασίας μας. Όταν μιλάμε για το άσυλο, για τη μετανάστευση, όταν μιλάμε για την ε, αστυνομική και δικαστική συνεργασία, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και όταν μιλάμε για οικονομική συνεργασία θα πρέπει να μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη μεν στους δε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι εργαζόμαστε βάσει των ίδιων αξιών, των ίδιων αρχών και ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στο σύστημα του άλλου, ό,τι το δικαστικό, για παράδειγμα, σύστημα. Να υπάρχει λοιπόν η ίδια βάση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αυτό είναι βασικό για την ιστορική αγορά. Σε όλους τους τομείς της πολιτικής λοιπόν είναι απαραίτητο να ξέρουμε ότι όλοι ξεκινάμε με την ίδια βάση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, αυτό που κάνει το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια είναι να καταρτήσει μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη δημοκρατία, το πρώτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί διαπιστώνουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλά νομικά μέσα για τους κανόνες, για παράδειγμα, κρατικών επιδοτήσεων, για τα περιβαλλοντικά πρότυπα, παραδείγματι, για τους κανόνες, για τα καρτέλα, αλλά δεν έχουμε αρκετά και ισχυρά μέσα για να υποστηρίξουμε και να υποστηλώσουμε αυτές τις αρχές και αξίες του άρθρου 2. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει συγκεκριμένα παραδείγματα για την απουσία σωστών μέσων. Αυτό έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ δύσκολε και ευαίσθητες, αν θέλετε, συζητήσει. Πέρσι τον Οκτώβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση της οποίας είχα την τιμή να είμαι υπεύθυνη για την κατάρτιση του. Και ο συνάδελφο, ο οποίο θα πάρει το λόγο αργότερα. Ο μηχανισμό λοιπόν που σχεδιάσαμε βασίζεται σε κάποιε αρχέ. Μία αρχή είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τη χάνουν ίσε μεταχειρήσει και θα πρέπει να αξιολογούνται με την ίδια ακριβώ βάση. Θα πρέπει να υπάρχει αντικειμενική αντικειμενικός τρόπος μέτρησης και α, αντικειμενική αξιολόγηση. Επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρχουν τρόποι αξιολόγηση σε διαρκέ και μόνιμο επίπεδο. Όχι κάθε φορά που υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Όχι, διαρκώ θα πρέπει να υπάρχει μια μέθοδο αξιολόγηση. Θα πρέπει να βασίζεται επίση σε τεκμήρια και να βασίζεται και στα υφιστάμενα μέσα. Δεν είναι δυνατόν να επανεφευρίσκουμε τον τροχό κάθε φορά. Και έχουμε και έτσι πολλά εργαλεία. των ετήσιων. Για παράδειγμα, κατάλογο επιδόσεων, το scoreboard, επίσης έχουμε το, την παρακολούθηση πλουραλισμού των μέσων ενημέρωση, έχουμε τη μηχανισμό συνεργασία και επαλήθευση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Έχουμε ήδη πολλά μέσα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Αν τα χρησιμοποιήσουμε όλα από κοινού με τον βέλτιστο τρόπο, θα έχουμε ένα πολύ καλό ετήσιο πλαίσιο για να παρακολουθούμε την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη, μια πάρα πολύ σημαντική αρχή και αυτό είναι ιδιαίτερα α, κέρια σημασία για τη σημερινή να, συζήτηση, είναι η συμπερίληψη των εθνικών κοινοβουλίων. Γιατί προφανώ όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν υπάρχει υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Το πώ ορίζουμε τι κοινέ αρχέ, τα κοινά πρότυπα, αποτελεί πραγματικά μια άσκηση η οποία θα πρέπει να γίνει από κοινού. Δεν θα είναι απλό. Και δεν είναι απλό, γιατί σίγουρα εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον έχουμε την ευκαιρία να βλεπόμαστε καθημερινά, να γίνεται αυτή η αντιπαράθεση καθημερινά, να κατανοούμε οι μεν του δε και να υπάρχει εμπιστοσύνη ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο όταν δεν υπάρχει καθημερινή επαφή. Και γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε και θα κλείσω λέγοντας αυτό, ότι αυτή η σημερινή εκδήλωση θα μπορούσε να γίνει μια ετήσια άσκηση, να υπάρχουν πιο πολλές ε, στιγμές ανταλλαγής απόψεων. Μία από τι απόψεις τι οποίε συζητήσαμε στο πλαίσιο της έκταση, την οποία μόλις ανέφερα είναι ότι κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να διορίσει έναν εισηγητή. Ένα άτομο, το άτομο επαφής μεταξύ του Εθνικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο ζήτημα της δημοκρατίας, κράτους δικαίου και θεμελιωδιών δικαιωμάτων. Αυτό θα ήταν πολύ πιο σωστό για την διευκόλυνση των σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ελπίζω ότι σήμερα οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα καταθέσουν καινούργιες προτάσεις για το πώς εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η συνεργασία και πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε κοινέ ε, αξίες και το πρωινό μας σήμερα το πρωί αυτό το γεύμα εργασία ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο. Ελπίζω να έχουμε και πιο πολλά τέτοια τέτοιες ευκαιρίες, γιατί αυτές οι μικρές ανεπίσημες συναντήσεις θεωρώ ότι είναι ενδεδειγμένε. Ε, για ε, ανταλλαγή απόψεων, πιο πολύ από δύο μεγάλε συνεδριάσει ενδεχομένω σε κάποιε περιπτώσει. Ε, σήμερα λοιπόν τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Έχουμε δύο πάνελ. Θα κάνουν εισαγωγέ ε, κάποιοι ομιλητέ. Έχουμε δύο ομιλητέ στο πρώτο πάνελ. Θα σα το παρουσιάσω σε λίγο. Θα μιλήσουν περίπου για 10 λεπτά και μετά θα έχουμε ένα γύρο ερώτα απαντήσεων. οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν απλά να σηκώσουν το χέρι και θα σας δίνω το λόγο. Τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να καταχωρήσουν το όνομά τους. Αν, αν παρακαλώ ζητήσετε από τους ε, υπεύθυνους να σημειώσουν το όνομά σας από τους κλητήρες, όπως ε, στη μέση εκεί της αίθουσας θα σημειώσουν το όνομά σας και θα μας φέρουν το σχετικό έντυπο. Άρα, το έντυπο για την πρώτη, το πρώτο ήμιση της συνεδρίασης είναι μπλε και κίτρινο για το δεύτερο ήμιση της συνεδρίασης για να δείτε το λόγο. Θα προσπαθήσω να το, να το κρατήσω όλο αυτό όσο πιο χαλαρό γίνεται, να δώσω το λόγο σε όσο πιο πολλούς γίνεται, αλλά και εσείς παρακαλώ δείξτε λίγο αυτοσυγκράτηση και λίγο αυτοέλεγχο σε ό,τι αφορά το Μέγεθο τη παρέμβασή σα. Δύο-τρία λεπτά νομίζω ότι αρκούν να πούμε τα αισιόδη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πάνελ και θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω από τον κύριο Φωντσέκα Μωρίγιο που κάθεται δίπλα μου να πάρει το λόγο που είναι ο αναπληρωτής ε, επικεφαλής της DG Just που είναι υπεύθυνη για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καλέσω τη συνέχεια του κύριου Βάνκλαφ Χάμποφ να πάρει το λόγο που είναι πρόεδρος της ε, Τσεχικής Γερουσίας της Σχετικής Επιτροπής για τα ζητήματα αυτά. Και μετά θα έχουμε γύρω ερωτοπαντήσεων. Έχετε το λόγο λοιπόν κύριε Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Ινβέλτ για την πρόσκληση. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του επικεφαλής μας, του κύριου Τίμερμανς, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει αυτή τη συζήτηση. Ήμασταν σιωπηλοί μάρτυρες ε, τη δεκαετία του 90 με τον πρόεδρο Ντελόρ ε, σε μια, στην πρώτη αυτή επαφή που είχαν ποτέ τα εθνικά κοινοβούλια με το Ευρωκοινοβούλιο. Βλέπω σήμερα πόσο έχει εξελιχθεί το πράγμα, πόσο συχνά συναντιόμαστε και μπορούμε να συζητάμε ε, την ε, δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, έχουμε κάνει ένα ψήφισμα που είναι αποτέλεσμα μιας εντυπωσιακή δουλειάς που έχετε κάνει εσείς, κυρία Ίντβελτ, ως εισηγήτρια. Ο πρώτος αντιπρόεδρος ε, Τίμερμανς και φυσικά ολόκληρη η Επιτροπή υποστηρίζει 100% της, ε, την ουσία του ψηφίσματος. Το βασικό είναι οι κοινέ μας αξίες να γίνουν σεβαστές και να εφαρμοστούν. Το θέμα είναι τώρα όχι, να δούμε τι θα γίνει με το άρθρο 2 της συνθήκης. Το βασικό θέμα της συζήτησης δεν είναι ο στόχος ο ίδιος όσο τα μέσα με τα οποία θα υλοποιήσουμε το στόχο. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν υποστηρίζει την ιδέα του ψηφίσματος να δημιουργήσουμε ένα διακοινοβουλευτικό διάλογο ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο. Ελπίζω πραγματικά η σημερινή ε, διακοινοβουλευτική συνεδρίαση να μην είναι μία μοναδική εκδήλωση και θα σταματήσει εκεί, αλλά να είναι η απαρχή ενός πραγματικού διαρθρωμένου διαλόγου ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια για το πώς θα εφαρμόσουμε, το πώς θα προωθήσουμε, το πώς θα στηρίξουμε τις κοινέ μας αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κατανοούμε με κοινό τρόπο ε, ως προς το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις κοινέ μας ε, αξίες και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορα σημαντικά θέματα, τα οποία αξίζει να συζητηθούν σε αυτή τη Διακοινοβουλευτική Επιτροπή, σε αυτόν τον διακοινοβουλευτικό διάλογο. Πρέπει να σκεφτούμε πριν το πώ θα εξασφαλίσουμε ότι οι ισχύουσε εκθέσει για την κατάσταση τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συζητώνται απλώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και κυρίω στα εθνικά κοινοβούλια δηλαδή η ιδέα του ψηφίσματος ότι τα ποικίλα δεδομένα και οι εκθέσεις που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν πιο προσπελάσιμα και σε εθνικό επίπεδο, φυσικά θα πρέπει να υποστηριχθεί. Υπάρχουν διάφοροι φορείς, το Συμβουλίο της Ευρώπης, η Επιτροπή της Βενετίας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, η ΦΡΑΚ, και μη κυβερνητικέ οργανώσει, προφανώ που ε, συνεισφέρουν στην παρακολούθηση τη δημοκρατία κράτου δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Αυτές οι εκθέσει και οι επίση αξίζει να τύχουν τη προσοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, η ΦΡΑ, παίζει ένα σημαντικό ρόλο ε, εξασφαλίζοντας αυτή την εύκολη πρόσβαση και την επισκόπηση όλης της πληροφορίας, όλων των εκθέσεων που αφορούν κάποια κράτη-μέλη, κάποια συγκεκριμένα θέματα. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί στο διακοινοβουλευτικό διάλογο θα είναι οι διάφορε εναλλακτικέ λύσει που έχουμε αυτή τη στιγμή για πιθανού νέου μηχανισμού για να προωθήσουμε τι κοινέ μα αξίε. Φυσικά, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα σύμφωνο για τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι μια βασική πρόταση επί της οποίας ε, καλό θα ήταν να ακούσουμε τις απόψεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Φυσικά υπάρχουν και άλλες ιδέες οι οποίες κυκλοφορούν και που αξίζει να ληφθούν υπόψη. Να υπενθυμίσω, Φερρυπίν, ότι το Συμβούλιο το 2014 δημιούργησε ένα διάλογο για το κράτος δικαίου ε, όπου συζητώνται όλα τα σχετικά θέματα. Πέρσι τον Νοέμβριο το Συμβούλιο αξιολόγησε το διάλογο και τα περισσότερα κράτη-μέλη τόνισαν τη σημασία εξασφάλισης της συνέχισης και ενίσχυσης αυτού του διαλόγου με πιο συχνές συζητήσεις που θα είναι προσανατολισμένε στα αποτελέσματα και καλύτερα διαρθρωμένε. Συμφώνησαν επίση ότι ο διάλογο αυτό για το κράτο δικαίου θα πρέπει να επαναξιολογηθεί στα τέλη του 2019 για να λάβουμε υπόψη τι δυνατότητε του να γίνει ο, αυτό το διάλογο να προκύψει και μία ε, έκθεση ομοτήμων που θα εκδίδεται κάθε χρόνο. Ο αντιπρόεδρο Τίμερμαν ε, τόνισε Επίση, και δεν θα σε εκπλήξει αυτό που θα πω, κυρία Ιντβελτ, ότι κάποιες ιδέες που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα ε, δημιουργούν ερωτηματικά και αμφιβολίες για μα την Κομισιόν, ειδικά για την ανάγκη και τη σκοπιμότητα αυτή τη ετήσια έκθεση και ενό κύκλου πολιτική για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που θα ετοιμάζει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Ο αντιπρόεδρος Τίμερ μας τόνισε ότι από πρακτική και πολιτική άποψη Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μια κοινή βάση για μια διαθεσμική συμφωνία μεταξύ όλων των διαφερομένων μερών που εμπλέκονται σε όλα αυτά τα θέματα. Η Κομισιόν θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση οι καλύτερες απόψη, η καλύτερη ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ισχύοντα μέσα και να μην τις, ε, να ε, υπάρξουν επικαλήσεις. Επίσης υπάρχουν ε, διάφορα και συμπληρωματικά μέσα για να προωθήσουμε και να στηρίξουμε τις κοινέ μας αξίες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω λοιπόν ότι η Κομισιόν έχει δημιουργήσει το πλαίσιο για το κράτος δικαίου, το οποίο εφαρμόζει ήδη στην περίπτωση της Πολωνίας. Δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι η Κομισιόν παίρνει πολύ στα σοβαρά το θέμα της προστασίας του κράτους δικαίου. Είναι ευγνώμων η Κομισιόν για την υποστήριξη που έχουμε λάβει από εσάς τους Ευρωβουλευτές. Επίσης άλλα υπάρχοντα εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να προωθήσουμε τις κοινέ μας αξίες. Φερρυπίν, η Κομισιόν ε, συνεχίζει να βοηθάει τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών δικαστικών συστημάτων με το ευρωπαϊκό ε, πίνακα αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη. Στην επόμενη σύνοδο θα έχουμε μια παρουσίαση του, αυτού του πίνακα αποτελεσμάτων του 2017 για την ε, δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη. Επίσης, για να είναι αποτελεσματική η χάρτα δικαιωμα... Ε, θεμελιωτών δικαιωμάτων, η Κομισιόν υποστηρίζει μια σειρά από ε, καταρχάς, την, το να συμμετέχουν όλοι οι επαγγελματίε του νομικού κλάδου σε αυτές τις διαδικασίες, οι δικαστές και οι εισαγγελίε. επίσης. δίνουμε σημασία στο να αυξήσουμε την κατανόηση των νομικών των ίδιων των ατόμων για το πώς μπορούν να σεβαστούν ε, οι ίδιοι ως άτομα καλύτερα τις α, θεμελιώδεις αξίες και να τις εφαρμόσουν. Προκειμένου να προωθήσουμε τις θεμελιώδεις α, αξίες, η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα ισχύοντα προγράμματα, τόσο ώστε να ενισχύσει τους φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κυβερνητικές οργανώσεις, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια αφύπνιση, μια συνειδητοποίηση για τη σημασία του θέματος σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό η Κομισιόν ενθαρρύνει την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να εργαστεί περισσότερο, τόσο ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητά από την κοινωνία των πολιτών αυτά τα θέματα και να καταλάβουμε καλύτερα πώς εξελίσσονται τα σχετικά πράγματα στην, στα κράτη-μέλη. Επίσης, θέλουμε η Ένωση να, προσ... να προσα να είναι συμβαλόμενο μέρο τη ε, σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται με πιο συνεπή τρόπο, πιο συνεκτικό τρόπο η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η Κομισιόν αξιολογεί συνεχώς το πώς τα ισχύοντα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια προ αυτή την κατεύθυνση. Είμαι πεπισμένο ότι μία διακοινοβουλευτική συζήτηση για τι διάφορε επιλογέ και θέματα θα βοηθήσει ούτω ώστε να να εντοπιστούν οι καλύτεροι τρόποι, ούτως ώστε να σημειώσουμε πρόοδο από κοινού. Κυρίε και κύριοι, για να ολοκληρώσω, θα πρέπει να μην υπάρχουν αμφιβολίες γύρω από τι κοινέ μα αξίε και θα πρέπει να υπάρχει συνένεση ε, γύρω από αυτά τα θέματα. Να προστατεύσουμε τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινή ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων και των ευρωπαϊκών και των εθνικών. Εθνικών φορέων και οργάνων. Χαίρομαι που σήμερα βλέπω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο δεσμεύονται να συνεργαστούν πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ε, έχουμε την λευκή βίβλο της Κομισιόν, όπου ε, αναφέρουμε ότι η δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια δέσμη αξιών που θα πρέπει να προωθηθούν από κοινού. Το μέλλον της Ευρώπης βασίζεται σε αυτέ τι αξίε. Ελπίζω αυτή η συνεισφορά του Αντιπροέδρου μα, κυρία Ίνθβελτ, να σας ικανοποιεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπω γνωρίζετε, εγώ πάντοτε θα πιέζω για περισσότερα και καλύτερα. Αυτό είναι το δικό μας το καθήκον. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χάμπλ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ο πλουραλισμός, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων νομίζω είναι ε, το σημαντικότερη περιουσία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως η ιστορία μας στην Ευρώπη μας διδάσκει ότι η δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένη στη Γερμανία, ε, στην Ιταλία, ε, ο κομμουνισμός στην πρώην Σοβιετική ε, Ένωση, τις πρώην χώρες της Ευρώπης που ανήκαν στο Σοβιετικό μπλοκ, μας έχει δείξει ότι η δημοκρατία χρειάζεται να περάσει από νέες διαδικασίες στις πρώην αυτές χώρες ε, κομμουνιστικές. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο μυστηριωδώς ε, προστατεύεται ε, από κάτι και το καθήκον του να φροντίσει κανείς τη δημοκρατία είναι φυσικά Είναι προφανώς ε, πρωταρχικός ρόλος κάθε χώρας και κάθε κυβέρνησης. Νομίζω ότι η δίψα για εξουσία είναι ένας πειρασμός ε, για τον άνθρωπο και ε, πολλές φορές υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τον καταμερισμό της εξουσίας θέλει κάποιο ενδεχομένως να έχει την εξουσία για πάντα. Νομίζω ότι είμαστε εδώ όμω για να υποστηρίξουμε ένα τον άλλον, να ε, βοηθήσουμε ένα τον άλλον υπό πολλέ έννοιε, να υποστηρίξουμε ένα τον άλλον ε, στην, ε, στον αγώνα, την προσπάθεια για μια καλή δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ σωστός αγώνας. Επιπλέον, εγώ είμαι του ιατρικού επαγγελματο και θα ήθελα μερικέ μερικές φορές χρησιμοποιώ παραδείγματα από το ανθρώπινο σώμα ε, όταν ένα από τα όργανα του ε, σώματος έχει κάποια δυσλειτουργία, ολόκληρο το σώμα υποφέρει. Επομένως, ε, αν δυσλειτουργεί η δημοκρατία σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό έμεσα ή άμεσα επηρεάζει αρνητικά τις υπόλοιπες χώρες. υπό τις ε, με τα δεδομένα αυτά λοιπόν, εγώ πρέπει να πω ότι έχω πραγματικά το μεγαλύτερο δυνατό συμβασμό για κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στο να ε, βρούμε ιδέες για να υποστηρίξουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον σε αυτόν τον αγώνα υπέρ της δημοκρατίας. Αυτό είναι εύκολο. Το να το πει κανείς. Το δυσκολότερο είναι πώς θα το κάνει κανείς με τρόπο που θα είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό. Το βλέπω κυρίως στη δική μου τη χώρα. Στη δική μου τη χώρα υπάρχει τεράστια εθνική ε, ευαισθησία σε σχέση με το τι μπορεί να θεωρηθεί εξωτερική ε, επιρροή βάσει των λόγων κάποιων πολιτικών ε, δημαγωγών που λένε ότι όλα αυτά προέρχονται από τις κακές Βρυξέλλες. Αν κάποιος προσπαθεί ε, να έχει πάνω από το δημοκρατικό κομμάτι της εξουσίας που θα του ανήκε ε, είναι μερικές φορές ε, ένας εχθρός. Είναι κάτι που πρέπει σε διεθνές επίπεδο να καταπολεμήσουμε. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Από νομική απόψεω έχουμε το άρθρο 7 ε, βεβαίω τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ε, θεωρείται μία προσφυγή τελευταία στιγμή ε, όταν η κατάσταση σε μία χώρα είναι πάρα πολύ κακή, ε, όταν υπάρχουν παραβιάσει τη ελευθερία των εκλογών, ε, τη ελευθερία έκφραση, τέτοιου είδου προβλήματα. Ε, ε, το, ο συνεχιζόμενος διάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προτείνει το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε προστιθέμενη αξία. Έχω τις αμφιβολίες μου. πρέπει να γίνει διάλογος και συζήτηση. Φυσικά αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ποτέ δεν, δεν κάνει κανείς αρκετό διάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, στην πράξη δεν είναι πάντοτε εύκολο να το κάνει κανείς. Ε, υπό τον όρο βεβαίως και οι δύο πλευρές ακούν ο ένας άλλον, ακούν η μία την άλλη ε, πραγματικά, ειλικρινά και δεν κάνουν συμναισθηματικές επικρίσεις ή δεν κατηγορούν ο ένα τον άλλον. Επίσης, ε, οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων μπορεί να έχουν κάποια προστιθέμενη αξία βέβαια μπορεί να είναι ένα και ένα παιχνίδι πολιτικών κατηγοριών, ένα πολιτικό παιχνίδι του τι κάνει η κυβέρνηση στη κάθε χώρα και ένα παιχνίδι που να ε, είναι ένα παιχνίδι παρέμβασης ε, στις εσωτερικές ε, υποθέσεις μιας χώρας. Μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων θα καταστήσει τον μηχανισμό βεβαίως αντιπαραγωγικό και ενδεχομένως επιβλαβή. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπάρχουν κάποιες αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές που είναι κοινέ για όλους, όμως υπάρχουν συγκεκριμένες παραδόσεις, ε, ε, μεθοδολογίες ε, που διαφέρουν μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Κάποια ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα κοινωνικά δικαιώματα για παράδειγμα, είναι αντικείμενο πολιτικής συζήτησης και πρέπει να αποφασίζονται από ε, τους πολιτικούς θεσμούς και όχι από τους εμπειρογνώμονες. Είναι λοιπόν δύσκολο για τους πολιτικούς θεσμούς να παραμείνουν αμερόληπτοι όταν πρέπει να κάνουν αξιολόγηση των επιδόσεων των άλλων. Εγώ προέρχομαι από ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον Οπότε θα μιλήσω κατά της δικής μου της κοινότητας κατά κάποιο τρόπο. Απλώς πιστεύω ότι το να επαφίεται κανείς τους εμπειρογνώμονες δεν είναι πάντοτε ε, η καλύτερη μέθοδος. Ε, υπάρχει μερικές φορές μια πολιτική προκατάληψη όσον αφορά κάποιες ιδέες. Ε, δεν κατηγορεί κανείς, ας πούμε, ένα χειρουργό για την απόφασή του να ε, ε, έχει χειρουργήσει ανάλογα με το αν είναι δεξιός ή αριστερός, για παράδειγμα. Ε, όμως όταν μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα, αυτό είναι μία πτυχή η οποία μπορεί να επισέρχεται. Το πρόβλημα που βλέπουμε με την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την εφαρμογή του κράτους δικαίου, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, και ούτω καθεξής. Ε, μερικές φορές εστιάζεται σε επίσημες πτυχές κατά πόσο ας πούμε ένας, ε, ένας νόμος έχει εγκριθεί ή όχι και λιγότερο κοιτάμε την, ε, το τι συμβαίνει στην πράξη και τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες αρχές συμπεριφέρονται. Η βελτίωση τώρα την κατάσταση, της κατάστασης σε σημαντικό βαθμό, εγώ νομίζω δυστυχώς ότι είναι λίγο εκτός των δυνατοτήτων των ε, ε, θεσμών της Ένωσης και των εμπειρογνωμόνων. Όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, φοβούμε πως είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαν τα εθνικά ε, κοινοβούλια να παρεμποδίσουν, να μπλοκάρουν το μηχανισμό ε, ώστε να αποφύγει μια χώρα να ξεφύγει από τη δημοκρατία. Να σκεφτώ ας πούμε την Αυστρία πριν από μερικά χρόνια όταν αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ε, ότι πρέπει από κοινού να υπερασπιστούμε την δημοκρατία στην Ευρώπη, το πρόβλημα δεν είναι τόσο ο Γιώργ Χάιντερ, δεν ήταν τόσο ο Γιώργ Χάιντερ, αλλά ε, το κόμμα του ε, και το κοινοβούλιο, ολόκληρο το κοινοβούλιο και το πόσο θα μπορούσε το κοινοβούλιο να βοηθήσει στην αποκατάσταση του προβλήματος. Δεν θέλω όμως να είμαι μόνο αρνητικός, θα θέλω να πω για μερικά θετικά. Ε, μπορώ να συστήσω την ε, εμπειρία που είχαμε εμείς με τη Γερουσία. Εγώ εκεί ανήκω. Η Γερουσία εκλέγεται διαφορετική χρονική στιγμή από το Κοινοβούλιο. Ε, το, η Γερουσία ασχολείται μόνο με την νομοθεσία, δεν ελέγχει την κυβέρνηση όπως το Κοινοβούλιο. είναι όμως εντελώς διαφορετικό το εκλογικό σύστημα για το ένα, για για την, την άλλη εκλογική διαδικασία. Και τα δύο σώματα όμως ε, δεν ε, είναι πολύ πιθανό να ε, κυριαρχείται από την ίδια συμμαχία ή από, την ίδια, από το ίδιο κόμμα. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και επηρεάζει το πώς λειτουργεί η χώρα επί καθημερινής βάσεως και αυτό είναι θεματοφύλακας του συνταγματικού, της συνταγματικής σταθερότητας γιατί χωρίς τη συγκατάθεση της γερουσίας δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή. Στη χώρα μας επίσης σημαντικές αποφάσεις ε, του Προέδρου της χώρας περνούν και από τη Γερουσία ε, και δεν έχει καμία σχέση με την πλειοψηφία που έχει κυβέρνηση ενδεχομένως ε, στο Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι περνάει ο χρόνος και ότι πρέπει να ολοκληρώσω. Θα ήθελα να προτείνω παρόλα αυτά την ιδέα της τακτικής παρακολούθησης, της κοινή παρακολούθησης ε, ε, των δικαστικών ε, διαδικασιών, του κόστους, των μακροχρόνιων διαδικασιών, των υποθέσεων που συζητούνται δημοσίως σε μια συγκεκριμένη χώρα, θα έλεγα ότι αυτό δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και μας δίνει κάποιες, κάποια στοιχεία και για το δικαστικό σύστημα της χώρας, αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση. Και επειδή έχω και κάποια εμπειρία από τη δική μου τη χώρα, κάτι τέτοιο έγινε και ε, για ε, δημόσιες υποθέσεις. Ε, ε, αν θέλει δηλαδή κανείς να διατηρήσει το επίπεδο της δημοκρατίας ή την ποιότητα της δημοκρατίας, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, πολύ πλούσια παρέμβαση. Uh, the Πριν ανοίξω το λόγο, δώσω το λόγο για συζήτηση, λίγες παρατηρήσεις ως συγγήτρια. Υπάρχει μια παρεξήγηση και δεν θα ήθελα να συνεχιστεί. Ειδικά, και θέλω να πω αυτό προς την Κομισιόν. Αυτό που δεν προτείνει το Κοινοβούλιο είναι ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων να παρακολουθεί τι κάνουν τα κρατημέλη και να προτείνει κυρώσεις. Η έκθεση θα συνταχθεί από την Κομισιόν, αλλά η διαδικασία θα εποπτεύεται από μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα διορίζεται εν μέρη από τα κράτη-μέλη και εν μέρη από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευρύτατη σύνθεση και θα κάνει συστάσεις. Δεν πρόκειται να αξιολογεί ή να τιμωρεί τα κράτη-μέλη. Και μια και τμήμα του μηχανισμού σημαντικό τμήμα είναι ο διάλογος και διακοινοβουλευτικός μάλιστα διάλογος, θα θέσουμε τα πρότυπα μαζί. Αναφερθήκατε νομίζω στο πανεπιστημιακό κόσμο. Υπάρχουν εκτεταμένοι μηχανισμοί για αξιολογήσεις, ε, αξιο... έκθεση ομοτήμων. Ε... Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα θα λειτουργεί και θα είναι ανθεκτικό. Ε, στο παρελθόν είπατε ότι πολλά αυταρχικά καθεστώτα δημιουργήθηκαν εκμεταλλευόμενα τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μηχανισμούς για να κρατήσουμε τις δημοκρατίες μας υγιείς. Αυτό ισχύει και για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Μερικέ φορέ θα πρέπει να ασκήσουμε αυτοκριτική. Δεν είναι και εύκολο, έτσι, γιατί είναι δυσάρεστο και πονάει. Αλλά είναι απαραίτητο. Και αυτό που είπατε και οι δύο και είναι από, ένα από τους βασικούς σκοπούς του συμφώνου που προτείνει το Κοινοβούλιο είναι η διαδικασία να αποπολιτικοποιηθεί. Γιατί μία διαφορά που έχω με τον κύριο Τίμερ μας και την Κομισιόν είναι ότι μα έχουμε το πλαίσιο του κράτους δικαίου και κοιτάξτε τι ωραία που λειτουργεί, γιατί το χρησιμοποιούμε κατά της Πολωνία. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί και τόσο καλά. Καταρχά, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και γιατί οι Πολωνοί θα αισθάνονται, Α, γιατί θελτεύετε εμά, γιατί μα κατηγορείτε, γιατί όχι τους άλλους. Κοιτάξτε του γείτονε. Και αυτοί κάνουν πράγματα που είναι λανθασμένα. Και εντάξει, κάπου έχουν δίκιο, έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ πιο εύκολα μερικές φορές για πολιτικούς λόγους επικεντρώνεται και κριτικάρει κάποιες χώρες και αυτό είναι εντελώ ανεπιθύμητο. Λοιπόν, αυτό το πολιτικό στοιχείο πρέπει να αφαιρεθεί και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο προτείνει ένα μηχανισμό που θα μεταχειρίζεται όλα τα κράτη-μέλη ισότιμα. Όλα τα κρατη θα αξιολογούνται πάνω στην ίδια βάση. Και θα έχουμε τα εξή δύο πλέον εκτήματα. Πρώτον, ότι δεν θα είναι μια πολιτική διαδικασία πλέον και οι κυβερνήσει δεν θα πρέπει να κρύβονται πίσω από αυτό το επιχείρημα πια και θα μα επιτρέψει να θέσουμε αυτά τα πρότυπα και να καθορίσουμε τα κριτήρια μαζί. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι 100%, αλλά αν είναι το αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας, θα είναι αποδεκτό σε όλους τελικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Επίσης αναφέρατε το εξής. Πώς ασχολούμαστε ή πώς αντιμετωπίζουμε κοινοβούλια ή ε, συγγνώμη, εθνικούς βουλευτές από χώρες που θεωρούνται ένοχες, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι τελικά, ακόμα και αν έχεις ουσιαστικές ε, διαφορές, μπορείς να κάτσεις, να συζητήσεις και να βρεις μια κοινή βάση. Και ναι, μπορούν τελικά να επιβληθούν κυρώσεις, αλλά είναι το τελευταίο μέσο, ε, όταν δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Όταν δεν εφαρμόζουμε ας πούμε, τους ε, περιβαλλοντικούς κανόνες ή τους ε, κανόνες για τον ανταγωνισμό, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, εφαρμόζουμε κυρώσεις, αλλά είναι πάντα η τελευταία λύση, η τελευταία έσχατη λύση. Έχω τώρα μία σειρά από άτομα που θέλουν να πάρουν τον λόγο. Ο κύριος Νίκος Πασκευόπουλος θα πάρει το λόγο πρώτα και συνεχεία ο κύριος Ενκόφσκι Βέτσεφ από την Πολωνία. Σε ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα για πρώτη φορά. Η χώρα μου ασπάζεται ασφαλώς τις αξίες της δημοκρατίας, των ε, ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και επίσης τους ε, ειδικότερους στόχους τους οποίους έχει τάξει αυτή η, Επιτροπή. Συμμετέχει βέβαια και στο πρόβλημα της απόστασης που υπάρχει καμιά φορά ανάμεσα στο επίπεδο των θεσμών και στο επίπεδο της πρακτικής εφαρμογής και πιστεύει ότι γι' αυτό χρειάζονται μηχανισμοί, ένας μηχανισμός παρακολούθησης και βεβαίως και ένας σύνδεσμος είτε αυτό μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των ε, κοινοβουλίων των ε, χωρών είτε αυτός ο σύνδεσμος θα είναι ένα όργανο, είτε θα είναι μονοπρόσωπος, είτε θα πρόκειται για μια μικρή κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω ακόμη στη διάθεσή μου πάντως, να εισφέρω και μία ακόμη πρόταση που πιστεύω ότι εμπίπτει στους στόχους της Επιτροπής αυτής. Ε, καταρχήν πλήρως τη σκέψη του Προέδρου Χέμπλ ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια περιουσία της Ευρώπης, θα έλεγα όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και της οικουμένης, της γης. Και πάντως είναι κυρίως ευρωπαϊκό έργο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο και από συμβολική και από πρακτική άποψη εάν η Ευρώπη θα αποκτούσε ένα μουσείο δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτό αν και πρόκειται για ευρωπαϊκό δημιούργημα. Ένα μουσείο θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ, όχι μόνο συμβολικά, αλλά και στη μελέτη και επίσης στην εκπαίδευση θεμάτων δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπάρχουν αντικείμενα στην ευρωπαϊκή ιστορία, είτε σύμβολα, είτε πρακτικά αντικείμενα τα οποία εξυπηρέτησαν τις λειτουργίες της δημοκρατίας και θα μπορούσαν να εκτεθούν. Η χώρα μου θα μπορούσε να προσφέρει ένα χώρο κοντά στην Ακρόπολη και τις αρχαιότητες της Αθήνας που να στεγάσει ένα τέτοιο μουσείο, αλλά πάντως δεν το βλέπει σαν ένα εθνικό πρόγραμμα. Γνωρίζει πολύ καλά ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, μπορώ να μνημονεύσω βέβαια ιδιαίτερα ίσως την Ιταλία, τη Γαλλία, αλλά όλες οπωσδήποτε οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εισφέρει στη δημιουργία της ε, δημοκρατίας με τη σημερινή της μορφή και όλες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού του μουσείου, να το διοικούν και γενικά να το αγκαλιάσουν. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Thank you very much. I think those... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν ε, πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά τα πράγματα που προτείνατε. Ο κ. Σεκόφσκι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ο διάλογος είναι πάντα σημαντικό στοιχείο. Ο διάλογος μεταξύ των κρατών μελών, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις Εθνικές ε, Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, με όλα τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί πρόκειται και για μια απόδειξη, αν θέλετε, του γεγονότος ότι η επιθυμία αυτή για τη συνδιαλλαγή με τα εθνικά κοινοβούλια είναι έντονη, είναι καλή η αρχή. Τώρα, το κατά πόσον το μοντέλο, κατά πόσον το σύστημα αυτό είναι το σωστό και το πιο ενδεδειγμένο, αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ε, διαμορφώνεται πάντα ως ε, συζήτηση μεταξύ εταίρων σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δραστηριοποιούνται. Το θέμα είναι και η εκπροσώπηση και η προάσπιση των ε, προβλημάτων και των ε, ανησυχιών των ε, πολιτών. Το θέμα λοιπόν τώρα είναι το monitoring, αυτός ο έλεγχος, η παρακολούθηση, η εποπτεία. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι ο τίτλος του μηχανισμού αυτού περιλαμβάνει και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου λοιπόν Στα πλαίσια του νομοθετικού πλαισίου, φυσικά. Αυτό σημαίνει κράτος δικαίου. Και τώρα προτείνεται ένας μηχανισμός ο, οποίος ξεπερνάει τα όρια του άρθρου 7 της συνθήκης. Μια κλειστή λεπτομερής διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη Θυμούμε με τον οποίο ελέγχεται κατά πόσο τα κράτη-μέλη πληρούν ή δεν πληρούν τι νομικέ προδιαγραφέ. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεπεράσει τα όρια τη σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητέ τη, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα αυτό ελέγχου. Και τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι υπέρ ε, φυσικά του ελέγχου και της καθοδήγησης, ασφαλώς, αλλά σε τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη είναι αυτά που παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν παρακολούθησης, αυτός ο μηχανισμός ελέγχου, ε, θεωρώ ότι είναι υπερβολικός, πάει υπερβολικά μακριά. Ένα εθνικό κοινοβούλιο για παράδειγμα. Αν υπάρχει αμφιβολία για ένα έγγραφο σε ό,τι αφορά ένα εθνικό κοινοβούλιο, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βγάζει κίτρινη κάρτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια, δυο, τρεις φορές στο κράτος μέλος Ποιος όμως ε, ελέγχει και καλεί να λογοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι γίνεται δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ένα εθνικό, ένα εθνικό κοινοβούλιο αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τηρεί τα άρθρα της συνθήκης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι πιο ενδεδειγμένο από τα εθνικά κοινοβούλια, ούτε είναι και καλύτερο από τα κράτη-μέλη ή πολίτες είναι η πιο σημαντική και με αυτού θα πρέπει να γίνει η συνδιαλλαγή, όχι με τέτοιο μηχανισμό όμως ελέγχου και παρακολούθησης. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Αν σας ε, καθησυχάζει, στην πρότασή μας περιλαμβάνεται και μια πρόταση να υπάρχει παρόμοιος μηχανισμός ελέγχου και για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Σόγκουρ τώρα έχει το λόγο. I'm sorry. Λυπάμαι, γιατί ακούγα στα ακουστικά την ερμηνεία. Θα μιλήσω ουγγρικά. Εμείς αυτό που θα θέλαμε θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλει να μπλεχτεί στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, δεν μπορεί στη συνέχεια να ενεργεί χωρίς νομική βάση από τις συνθήκες. Δεν μπορούμε απλά να αποφασίσουμε ότι θέλουμε ένα τέτοιο μηχανισμό και στη Ρουμανία τα γεγονότα της εβδομάδας αυτής όλοι οι υπουργοί εξωτερικών υποθέσεων, η πρωθυπουργό κτλ. Κάναν δηλώσει και τι βλέπουμε στην ε, πράξη. Ότι όταν η κατάσταση επιδεινώνεται, υπάρχουν, ε, για παράδειγμα, ε, νομοθεσίες για τις ε, μειονότητες σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους, τη γλώσσα τους, την εκπαίδευσή τους, για να ξέρουν οι γονείς γιατί στέλνουν τα παιδιά τους σε ειδικά σχολεία. Αν, λοιπόν, το θέμα δεν είναι η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία αν γίνει δεκτό αυτό ως αρχή, Υπάρχουν λοιπόν κανόνες σε ό,τι αφορά τις μειονότητες, όπως στη Σλοβακία για παράδειγμα. Και σε ένα μόνιμο επίπεδο υπάρχει επίθεση κατά των α, μειονοτήτων και κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν από την κυβέρνηση για τις μειονοτητές. Για να δούμε λοιπόν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα πραγματικά να γίνουν σεβαστές ε, οι συνθήκες. Thank you very much. Next on my list, Mr. Επόμενος, παρακαλώ, ο κύριος Ντίρκα από τη Ρουμανία. probably just massacred your last name. Sorry about that. Ε, don't worry. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριοι και κύριες ε, βουλευτές, με μεγάλη τιμή εκπροσωπώ εδώ το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ποιο είναι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτό. Από την αρχή θα ήθελα να σας πω ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα μπορεί να μας ανοίξει την πόρτα για αυξημένες ευθύνες σε ένα πολύ περιπλοκό τομέα. Ε, ένα τομέα που μέχρι τώρα ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών κρατών, των κρατών δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας ε, στεναρός μηχανισμός έχει διάφορα εργαλεία που μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές. Θα ήθελα να μιλήσω για το άρθρο 4 παράγραφος 2 της συνθήκης. Θα ήθελα να μιλήσω και για τα πολιτικά κριτήρια, για το πολιτικό κομμάτι μάλλον της, των κριτηρίων της Κοπενχάγης, κυρίως το άρθρο 6. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο άρθρα. Φυσικά, υπάρχουν ε, οι κανόνες από τη μία, οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Μερικές φορές υπάρχουν και κάποιες διολυστήσεις σε εθνικό επίπεδο. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν μια κοινή προσπάθεια, ούτως ώστε να προστατεύσουμε περισσότερο τα κρατη μελη πρεπει να κανουν μια κοινη προσπαθεια ωστε να προστατευσουμε περισσοτερο τα συμφεροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Το κράτος δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να, να λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις αρχές και θα πρέπει να είναι στη βάση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές. Τα κράτη-μέλη ε, δουλεύουν με συνενετικό τρόπο και ο μηχανισμός ελέγχου της δημοκρασίας και του κράτους δικαίου είναι μια προτεραιότητα ούτω ώστε να δημιουργηθεί μια μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική που θα μπορούσε να εξασφαλίζει μια καλή λειτουργία του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει οι πολιτικές εξελίξεις ε, στα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους ένα τέτοιο μηχανισμό που ελπίζω να δημιουργηθεί κάποια στιγμή αυτός ο μηχανισμός. Και να υπάρχουν και κυρώσεις για όλα τα κράτη-μέλη που θα είναι στην καρδιά μιας τέτοιας πολιτικής. Όπως ξέρετε, στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μηχανισμό συνεργασίας και επαλήθευσης που έχει αποδείξει ότι λειτουργεί, ήταν αποτελεσματικό εργαλείο και μας επέτρεψε να σεβαστούμε καλύτερα το κράτος δικαίου. Να υπάρχει ένα τέτοιο μηχανισμό για όλα τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ε, συνθήκες. Να σας ότι η Ρουμανία επικύρωσε και σεβάστηκε όλα τα κριτήρια αυτού του μηχανισμού επαλήθευσης. Πιστεύουμε ότι αυτός ο μηχανισμός τώρα θα πρέπει να αφήσει λιγάκι ήσυχη τη Ρουμανία γιατί κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Διντιέ Μαγί, από τη Γαλλία είναι επόμενο στη λίστα μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να επικροτήσω την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο αγαθό και το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε και παράλληλα το πιο ευάλωτο. Όλες οι πρωτοβουλίες λοιπόν που έχουν σκοπό να ε, διατηρήσουν ε, την ε, δημοκρατία για τους πολίτες μας πρέπει να επικροτείται. Αυτό αναφερόταν βέβαια και στα προκαταρτικά ε, σχόλια. Πάρα πολλέ πρωτοβουλίε λαμβάνει η χώρα ε, στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια υπηρεσία που δημιουργείται, όλα αυτά που πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να υπάρχει βέβαια και σωστό συντονισμό των πρωτοβουλειών, να μην υπάρχουν ε, αλληλοεπικαλύψει ώστε οι πολίτες μας να μπορούν να καταλάβουν καλά το τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε, σχέση, σε συνεργασία με τα ε, Εθνικά Κοινοβούλια. Σήμερα, και συμφωνούμε με αυτή τη διαπίστωση, υπάρχει στην Ευρώπη, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, ε, σοβαρή παραβίαση της δημοκρατίας, ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών και στο μεγαλύτερο τμήμα των κρατών μελών ε, μπορεί να σημειωθεί πρόοδος ε, και στη Γαλλία μπορώ να πω όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την ελευθερία των, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την ισότητα ανδρών και γυναικών, το σεβασμό των μειονοτήτων, ε, την ε, ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίες και αναφέρομαι κυρίως στο ζήτημα των μεταναστών. Η επαγρύπνηση λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητη και οποιοδήποτε μηχανισμός επιτρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υποστηριχθεί. Όμως η επαγρύπνηση δεν επαρκεί. Πρέπει ε, όταν χρειάζεται να μπορούμε να δημιουργήσουμε αποτελεσματικές διαδικασίες, δεσμευτικές διαδικασίες, ε, αφού θα έχουμε εξαντλήσει όλη τη δυνατότητα διαλόγου, ότι το άρθρο 7 των συνθήκων να μην είναι μία μνήα απλή, αλλά να εφαρμόζεται αποτελεσματικά όταν υπάρξει ανάγκη. Είμαστε λοιπόν υπέρ ενός μηχανισμού ολοκληρωμένου, και πιστεύω ότι η συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και σε άλλους τομείς, νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητη. Εμείς θα είμαστε προσεκτικοί και μας ενδιαφέρει η επεξεργασία του μηχανισμού αυτού που ε, θέλετε να προτείνετε. Ο διάλογος, ο διάλογος πάντοτε είναι καλός, αλλά μετά το διάλογο κάποια στιγμή πρέπει στην πράξη τα θεμελιώδη δικαιώματα να γίνονται σεβαστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ντάρλεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, συμφωνώ με τον συνάδελφο γερουσιαστή Didier Μαρή ε, και για να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε προηγουμένω, κυρία Πρόεδρο, όσον αφορά τη χρησιμότητα και τη σημασία του να μπορούμε ε, να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει εκλεγεί από του Ευρωπαίου πολίτε και τα εθνικά κοινοβούλια να συνεργάζονται, γιατί από ό,τι κατάλαβα από τι παρεμβάσει των ΜΕΝ και των ΔΕ έχουμε την ίδια πεποίθηση, ότι η προάσπιση των ε, αξιών ε, που μας ε, ε, φέρνουν κοντά ε, στον έναν τον, τον έναν στον άλλον είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι αξίες όπως και η ενιαία αγορά, όσο και οι οικονομικές συναλλαγές, αλλά και οι κοινέ αξίες μας. Και πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε ότι ο σεβασμός των διατάξεων που αφορούν την ελευθερία ε, κυκλοφορίας των κεφαλαίων και ελευθερία των, στο, στις αγορές να ε, ισχύει για όλους, ε, ε, δεν Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να αντιβαίνει στην προάσπιση των αξιών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε ε, νομίζω ότι γι' αυτό γίνεται, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία ε, που είναι αντικείμενο τόσων πολλών συζητήσεων για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να προχωρήσουμε περαιτέρω γιατί τα νομοθετικά εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας ε, μας δείχνουν ότι δεν είναι αποτελεσματικά ε, δεν είναι στο επίπεδο του μηχανισμού οικονομικής σταθερότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ενέκρινε ε, αυτόν τον μηχανισμό και χαιρετίζω την προδραστική διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, εφαρμογή του μηχανισμού αυτού. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω και από τα Εθνικά Κοινοβούλια να μην θεωρήσουν ότι αυτή η παρακολούθηση, η εποπτεία είναι κάτι το αρνητικό. Ε, είναι ένας τρόπος να διατηρήσουμε τη ζωτικότητα της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης, χωρίς την οποία θα εξαφανιστεί. Ε, πρέπει να το δείτε λοιπόν επικοδομητικά. Ε, υπάρχει ένα θέμα λοιπόν ε, και με την χρονική ε, στιγμή είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα. Είχαμε πει το 2005 ήδη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ότι το 2020 θα το ξαναδούμε, αλλά όχι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να αναλάβουμε όλοι τώρα τις ευθύνε μας και να εργαστούμε χωρίς να λέμε ότι είναι ένα θεσμός, ένα κοινοβούλιο εναντίον σε ένα άλλο. Δεν πρόκειται καθόλου περί αυτού πρόκειται για το σεβασμό των ε, αξιών ε, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που πρέπει να γίνεται παντού με τον ίδιο τρόπο και όταν υπάρχουν παραβιάσεις ε, ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι δυνατόν να το παραγνωρίζουμε και να δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιους να μην τα σέβονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνιο Φελίπε από την Πορτογαλία είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Σε ό,τι αφορά θέματα αρχής, θα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν σε δημοκρατικές χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα όμως είναι τι γίνεται όταν περνάμε στη φάση της υλοποίησης, της εφαρμογής. Εδώ αντιμετωπίζουμε δύο προβλήματα θεωρώ. Καταρχάς, ποιος θα ορίσει τις καλύτερες ε, δομές για την εφαρμογή των αρχών. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Αν όλοι συμφωνήσουμε για το εκλογικό σύστημα, εγώ μπορώ να πω ότι το δικό μου εκλογικό σύστημα είναι καλύτερο και πιο δίκαιο από το δικό σας. Ποιος θα αποφασίσει τελικά ποιο είναι το καλύτερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε πιστεύω ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο για όλα τα κρατή μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μετά ανακύπτει το ερώτημα του ποιο θα είναι αυτό που θα το αποφασίσει. Δεύτερο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά από την αναγνώριση των, από πλευρά των πολιτών της ε, δημοκρατικής νομιμότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι πολίτες δεν έχουν την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μοντέλο δημοκρατίας. Θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο τους ε, επιβάλλεται εκ των άνωθεν και αναγκάζεται να το τηρήσουν και να το εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Αυτή η έλλειψη λοιπόν αναγνώριση ε, της ε, δημοκρατικής νομιμοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την επιβολή κυρώσεων στα κράτη-μέλη. Για να τελειοποιήσουμε λοιπόν τη δημοκρατία, θεωρώ ότι θα πρέπει ενδεχομένω να συμμετέχουμε πιο έντονα. Θέλουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμμετέχουν και φυσικά τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά δεν πιστεύω ότι το να απειλούμε με κυρώσεις αποτελεί το σωστό τρόπο να προχωρήσουμε. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε τον κόσμο, γιατί αυτό μοιραία θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και του πολίτη. Είναι φυσικά στη θεωρία όλα τα κράτη-μέλη ίσα. Ξέρουμε όμως στην πράξη αυτό δεν ισχύει και ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι να οξυνθούν οι υφιστάμενες συντάσεις μεταξύ των διαφορών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος ε, του κράτους μέλους και την σφαίρα επιρροής του, αυτή η ισότητα μεταξύ των κρατών μελών Μπορεί να ισχύει επί τη αρχή, αλλά απέχει παρασάγκα από το να βρίσκεται στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Δεν θα απαντήσω τώρα, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε αυτέ οι συζητήσει και εμεί τι έχουμε συζητήσει επί μακρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πολλά τα θέματα τα οποία τίθεται. Η κυρία Στίνα Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Στην Ολλανδία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε ότι η δημοκρατία δεν, αφορά, δεν είναι μόνο το θέμα των εκλογών. Είναι το πώς θα ανακάσουν οι πολίτες να λογοδοτήσουν ε, οι κυβερνήσεις τους. Θα ανακάσουν τις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν και να το κάνουν κάθε μέρα. Και το θέμα είναι πώς αυτές οι πρωτοβουλίες των ε, πολιτών συνδέονται με αυτό το μηχανισμό. Πώς θα εμπλέξουμε τους πολίτες σε αυτό το μηχανισμό, πώς θα τους ε, επιτρέψουμε να μιλήσουν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και ακόμα πιο σημαντικό πώς θα συντονίσουμε τις προσπάθειες των πολιτών και των κινημάτων των πολιτών ε, χωρίς το πρόσκομα των εθνικών συνόρων, τόσο ώστε να αισθανθούν αλληλεγγύοι, ούτω ώστε να είναι ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτε για θέματα πολύ σημαντικά, τα δικαιώματα των γυναικών, των μειονοτήτων, των ΛΟΑΔΑ. Πώς θα θεωρήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι αυτός ο μηχανισμός του αφορά. Όχι μόνο να διαβάζουν τις εκθέσεις δηλαδή των ε, εμπειρογνωμόνων από τις αιτήσει συνεδριάσει τους δηλαδή, αλλά πώ θα του εμπλέξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω συμμετάσχει και φυσικά έχω υποστηρίξει στεναρά αυτή την έκθεση τη Σόφη Ιντφέλτ. Και με τα ταύτα μπορώ να σας πω ότι αυτή την ε, συνάντηση τη θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι χρήσιμη γιατί ξεκινάει και φυσικά χωρίς κανένα, χωρίς να γίνει τίποτα έξωθεν, βλέπω ότι αρχίζουν να δημιουργούνται παρεξηγήσεις ήδη. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, τι μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο μηχανισμός, και ας με διορθώσει η Σόφια αν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε και για να, για να αξιολογήσουμε με κριτικό τρόπο όλες τις μεθόδους που χρησιμοποίησαμε μέχρι στιγμής, ούτω ώστε να προωθήσουμε το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω να ξεχάσουμε τους ισχύοντες μηχανισμούς, όχι, να τους κρατήσουμε, αλλά υπάρχουν, υπάρχει μια προστιθέμενη αξία σε αυτό το μηχανισμό. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ποιοτικό άλμα που κάνουμε με αυτό το μηχανισμό. Και μάλιστα θα έλεγα δύο ποιοτικά άλματα τα οποία μάλιστα εν μέρη περιγράφηκαν. Λοιπόν, το πρώτο άλμα είναι ότι είναι ένας μόνιμος μηχανισμός που δεν έχει σκοπό να παρέμβει απλώς για να διορθώσει μια ζημιά, αλλά να προλάβει μια ζημιά. Επομένως, αυτή την ιδέα, με τις που έχουν άλλοι μηχανισμοί, εδώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζεται πάρα πολύ σε μια ανεξαρτησία και στην αμεροληψία ας πούμε των εμπειρογνωμόνων. Μιλάμε για εμπειρογνώμονες που δεν είναι πολιτικοί, που είναι ανεξάρτητοι από την πολιτική. Ψάχνουμε δηλαδή σε αυτό το σώμα εμπειρογνωμόνων να βρούμε άτομα για να συμμετάσχουν, τα οποία θα είναι αμερόληπτα ε, και θα εκφράσουν μια πλειάδα απόψεων. Και θα μας βοηθήσει επίσης να ξεπεράσουμε αυτήν την ιδέα της τιμωρίας. Τιμωρίες που επιβάλλουν τα θεσμικά όργανα μερικές φορές. Μην ξεχνάτε ότι και τα ίδια τα θεσμικά όργανα είναι υπό επιτήρηση. Και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κάτω τη γνώμη μου, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν ίσως στα χέρια τους αρκετούς δείχτες, αρκετούς, αρκετές παραμέτρους. Ε, νομίζω ότι και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να τα εξετάζουμε σε αυτή την ε, έκθεση και να έχουμε και τις α, παραμέτρους και τους δείκτες. Λοιπόν, και μια προσωπική παρατήρηση για, τον, ε, για τη λέξη, για την φράση, αν θέλετε, κοινέ αξίε. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν ήρθα από την αρχή, γιατί θα το είχα πει αυτό από την αρχή. Φυσικά οι αξίε υπάρχουν στι συνθήκε. Έτσι, αναφέρονται στι συνθήκε. Είναι όμως μία λέξη που δημιουργεί αφησιμίες. γιατί συχνά οι αξίες είναι κάτι το πολύ υποκειμενικό. Συνδέεται με, το, με την κουλτούρα, με τον πολιτισμό. Συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε παραδόσεις. Εγώ, αν ξανάγραφα τι συνθήκες, θα προτιμούσα να μιλάμε για κανονιστικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεμέλια τα νομοθετικά. Και σε αυτό βασίζεται η έκθεση της Σοφή. Αυτό είναι το κοινό μας πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες, το δίκαιο, δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Δεν είναι υποκειμενικό το δίκαιο. Υπάρχουν στη συνθήκη. Δεν είναι αντικείμενο διαλόγου. Είμαστε υπέρ, είμαστε κατά. Γιατί πέραν του ότι αναφέρονται σε συγκεκριμένα άρθρα των συνθήκων, υπάρχουν και στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει την ίδια αξία. Η χάρτα έχει την ίδια αξία με τις συνθήκες. Ο Πολωνός συνάδελφος μας ρώτησε ποιο είναι το μοντέλο στο οποίο αναφερόμαστε. Το θέμα δεν είναι το μοντέλο. Το, θέμα είναι τα συγκεκριμένα άρθρα της συνθήκης και των θεμελιωδών και των συνθήκων. Συγγνώμη. Όσο περισσότερο συζητάμε, τόσο περισσότερο ξεκαθαρίζουμε τα θέματα αυτά. Και τόσο περισσότερο πλησιάζουν οι θέση μας. Εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν δημιουργεί γεννά πάρα, πολλούς, πάρα πολλές αμφιβολίες για αυτό το μηχανισμό. Και η ίδια στο μυαλό της έχει και προκαλεί. Ε, δεν είναι ένας ακόμα μηχανισμός, είναι ο μηχανισμός. Ο κύριος Μικολάσιτς από την Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. κύριε και κύριοι. Χαίρομαι πραγματικά που συμμετέχω σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική συνεδρίαση. Εκπροσωπώ το, τη γερουσία της Πολωνικής Δημοκρατίας και κυρίως την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της ε, αναφορές και το κράτος δικαίου. Ως Επιτροπή ασφαλώς ε, συμμετέχουμε με τα ζητήματα αυτά, στα ζητήματα αυτά και συνεργαζόμαστε με εκπροσώπους των πολιτών και τα θέματα λοιπόν αυτά θα πρέπει να θίξουμε. Τα θέματα τα οποία αναφέρονται και στην ημερήσια διάταξη για το διάλογο τώρα. Αυτός ο διάλογος είναι πραγματικά απαραίτητος και αποτελεί και μία από τις αρχές του κράτους δικαίου σε ένα κράτος το οποίο υπάρχουν και ισχύουν τα θεμελιώδη ανθρωπινά δικαιώματα. Αλλά μιλάμε για κυρίαρχα κράτη τα οποία ανταλλάσσουν αντικειμενικά τις απόψεις τους. Εγώ πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενδεχομένω θα πηγαίνουν και λίγο υπερβολικά μακριά σε ό,τι αφορά δηλαδή θέματα ε, Παραβίαση της ε, επικυριαρχίας των κρατών μελών και της αξιοπιστίας, ε, ενδεχομένως από πλευράς των πολιστών, της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων. Ο αμοιβαίος σεβασμός έναντι των κρατών μελών. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η εμπιστοσύνη όμως ασφαλώς προϋποθέτει και αναγνώριση των ε, αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο εθνικών κρατών μελών. Φυσικά θέλουμε να συνεχίσουμε το διάλογο. Και όπως είπατε εισαγωγικά, θα πρέπει να υπάρχει αμερόληπτη αξιολόγηση των δράσεων των άλλων παραγόντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Αζουμπάλης από τη Λιτουανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή, το φωτοκείμενο το οποίο μας ε, λάβαμε. Να σχολιάσω το άρθρο υπαριθμών 8 σε ό,τι αφορά τα πάνελ των εμπειρογνωμόνων, expert panel. Φαίνεται... ότι η ερμηνεία των αξιών και των ε, θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι 100% στα χέρια των δικηγόρων. Και δικηγόροι, ξέρετε, πολλές φορές δεν περιγράφονται με ωραίους όρους. Αυτά τώρα φυσικά είναι και ιστορικά ζητήματα. στον κατάλογο των εμπρεγνωμόνων, των αποκαλούμενων εμπειρογνωμόνων, δεν βλέπω να υπάρχουν εκπρόσωποι από άλλους επαγγελματικού κλάδους. Μόνο νομικού ε, και δικηγόρου. Μόνο στου δικηγόρου βασίζεται και στον νόμο βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο οι δικηγόροι και οι νομικοί έχουν άποψη. Αμφιβάλλω, πραγματικά. Πέραν αυτών, ε, έχω φυσικά απόλυτο σεβασμό προς ε, τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΣΑ. Πρόκειται για πολύ σπουδαίους ε, διεθνείς οργανισμούς, αλλά συνδέονται με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ναι, σε περίπτωση που είναι μέλη των οργανώσεων αυτών. Αλλά για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ποιο μπορεί να αποφασίσει ποιο εμπειρογνώμονα ε, θα συμμετέχει στο πάνελ των εμπειρογνώμονων, η Προεδρία, ο Γενικό Γραμματέα. Το ίδιο ισχύει και για τα Ηνωμένα Έθνη. Ποιο παίρνει τι αποφάσει, ε, η Γενική Γραμματή, άλλοι. Κάθε οργάνωση έχει τα καθήκοντά της. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει κάτι με τι ε, υποχρεώσει των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη έχουν υποχρεώσει έναντι των οργανώσεων. Αν δεν τι στηρίσουν, τότε μάλιστα μπορούν να λάβουν μέτρα οι οργανώσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων με τα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Εθνικό Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει έναν εμπειρογνώμονα και κοιτώντας τι προτείνει η Ευρωπαϊκή, Επιτρο... η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπάρχουν κριτήρια για το ποιο εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό προτείνεται. Μα φαίνεται λοιπόν ότι η πρόταση αυτή θα περιορίσει τις αρμοδιότητες των Ευρωπαίων πολιτικών να λαμβάνουν αποφάσεις και θα αντίθεται εξωτερικά στις επωνομαζόμενες ανεξάρτητες οργανώσεις οι αποφάσεις αυτές, η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, στο τέλος της συζήτησης θα κάνω κάποιες διευκρινήσεις για τον ρόλο των πάνελ των εμπειρογνωμόνων και σε ό,τι αφορά για τις προτάσεις, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις. Κύριε Φωστόρχη, στη λόγο. Σα äh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε εισαγωγικά ότι το άρθρο 2 είναι σημαντικό και είπατε ότι εκεί κατοχυρώνονται οι αρχές. Ε. Είπατε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε αξίες και αρχές και μετά είπατε ότι θα πρέπει να οριστούν αυτέ οι αξίε γιατί ο καθένα καταλαβαίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό λοιπόν ισχύει. Εσεί καταλαβαίνετε κάτι διαφορετικό με τον όρο δικαιοσύνη από ότι εγώ ή από ότι πολλοί άλλοι εκπρόσωποι. Για εσάς η άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Για εσά, η άμβλωση είναι άλλου, η ενός θανατος ενό όντους. Δεν θέλω να παρέμβω στι δικέ σα απόψει, αλλά αυτό που ονομάζετε εσεί ω ε, ως αξία και αρχή ε, δεν το σπάσονται άλλοι. και θέλετε λοιπόν αυτό το μηχανισμό για τα πράγματα τα οποία ερμηνεύονται και δεν είναι σαφή. Αυτές τις αξίες λοιπόν θέλετε τώρα σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα κρατημέλη να τα εφαρμόσετε, να τα επιβάλλετε. Να παρακάμψετε τις αρχές που υπάρχουν τα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέλετε λοιπόν να βγάλετε ένα πολιτικό πάνελ εμπειρογνωμόνων για τις αξίες που έχετε εσείς και πολλοί δεν συμφωνούν με αυτέ, Δεν τι επιβάλλετε. Το είπε ένα από του Γάλλου συναδέλφου προηγουμένω ότι η εποπτεία δεν είναι κάτι αρνητικό, είναι ε, μια ένδειξη ζωντάνια. Θέλετε λοιπόν να παρακολουθείτε τα κράτη-μέλη που δεν ασπάζονται τι αρχέ σα και μετά λέμε ότι είναι ένδειξη ζωντάνιασμα και η Σοβιετική Ένωση λοιπόν και η Βόρεια Κορέα είναι πάρα πολύ ζωντανέ ε, χώρε. Για σκεφτείτε λοιπόν τι θα συνέβαινε αν οι αρχέ οι οποίε είναι δικέ σα αξίε και δεν αμφισβητώ αυτό, δικέ σα είναι, τι κάνετε ό,τι θέλετε. Και όταν λέω εσά είναι δικέ σα αξίε, εννοώ ότι και μια μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασπάζεται ε, τι ε, αξίε σα ότι ο γάμος, για παράδειγμα, είναι ασθένεια, προκαλεί νόσο. Αυτές είναι οι δικές σας αξίες, τις οποίες τις ασπάζετε, τις ασπάζετε και με μια μεγάλη πλειονότητα εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σας ασπάζετε όμως μεγάλη πλειοψηφία των, ε, των ε, εθνικών βουλών. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση από πλευρά ε, των Ευρωπαϊκών κρατών, γιατί πολύ απλά δεν ασπάζονται τις αξίες σας. Κυρία Φωνστόρχ, λέει η Πρόεδρος, υπάρχουν κάποιες ε, εικασίες επί των οποίων δεν συμφωνώ πολύ απλά. Και να σας πω και την αλήθεια, είναι λίγο σαν γελιογραφία αυτό που παρουσιάζεται. Καρικατούρα. Η έκταση υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μία μειοψηφία η οποία δεν συμφώνησε. Αλλά να μα λέτε τώρα Σοβιετική Ένωση και Βόρεια Κορέα, νομίζω ότι κάπω υπερβάλλεται. Ο κύριος Βίλτερ από την Ολλανδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά και χαίρομαι που βρισκόμαι εδώ και χαίρομαι που έχουμε και κάποιους συναδέλφου από την Πολωνία μαζί μας και από την ε, Ουγγαρία. Μπορούμε να μιλήσουμε για την πρόταση και για την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ έχω να θέσω το εξή και θα ήθελα να απευθυνθώ κατευθείαν στους συναδέλφους από την Πολωνία και την... Ε, στη χώρα μου την Ολλανδία επικρατεί σκεπτικισμός ε, μεταξύ κάποιων ε, συμπατριωτών μου. Κάποιοι λένε ότι πήγε πάρα πολύ γρήγορα η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέθηκαν πάρα πολλές χώρες οι οποίες δεν ασπάζονται τις ίδιες αξίες. Και αναρωτιούνται αυτοί οι πολίτες τι χώρες έχουν πλέον προσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ε, έχουν τις ίδιες αξίες και η Ολλανδική νομολογία, τα δικαστήρια ε, έγραψαν ε, μια επιστολή προς το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη στην Πολωνία και αποφάνθηκαν οι δικοί μας δικαστές ότι δεν πάνε τα καλά τα πράγματα με την δικαιοσύνη στην Πολωνία. Πώς θα εξηγήσω λοιπόν, σας ερωτώ, στο εκλογικό μου κοινό που εν μέρει είναι ευρωσκεπτικιστές, το τι συμβαίνει στην Πολωνία. Πώ θα τα εξηγήσω και πώ θα τα βελτιώσουμε όλα αυτά. Πείτε μου λοιπόν τι να απαντήσω στον κόσμο για να υπάρχει υποστήριξη και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και προ την Πολωνία. Okay, thank you very much. ευχαριστώ πολύ. Τρει ακόμα θα ακούσουμε στο πρώτο αυτό πάνελ. Τρία ακόμα άτομα και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Χάμπερ και στον κύριο Μολίγη για να κάνουν τα καλλιτικά του σχόλια. Δύο αιτήματα από εθνικά κοινοβούλια. Ο κύριος Μποντρή από το Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ κύρια ε, Πρόεδρε. Όπως είπαν πολλοί ως τώρα, είναι πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή που αναλάβατε, γιατί εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι το ζήτημα ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ε, και του κράτους δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα για να τα αφήσουμε μόνο στις κυβερνήσεις. Πρέπει λοιπόν και τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν ε, και να υπάρξει διάλογος μεταξύ των διαφόρων εκπροσώπων του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όμως, και εδώ θα σας πω ήδη κάποια πρώτα σχόλια σε σχέση με αυτό, η επισημοποίηση του διαλόγου αυτού μέσω μιας ε, ε, διεθνούς συμφωνίας ε, δεν θα μπορέσει να αποτελέσει το σημείο αφετηρίας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιασμοί ακόμη και εντός αυτής της αίθουσα, και είναι σίγουρο ότι εφόσον υπάρχουν εδώ θα τις δούμε και σε επίπεδο Υπουργείου, συγγνώμη, Συμβουλίου Υπουργών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην εστιάσουμε πάρα πολύ ε, στην δημιουργία ενός ε, επισήμου πλαισίου που μερικές φορές ε, δεν, δεν επιφέρει αυτήν την προστιθέμενη αξία που θα θέλαμε για το άρθρο 13 για παράδειγμα. Δύο χρόνια μιλήσαμε για τους κανόνες λειτουργίας αυτής της συνεργασίας εθνικών και ευρωπαίων βουλευτών και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξει πουθενά. Είναι σημαντικό λοιπόν πολλές φορές να συναντιόμαστε με πολύ συγκεκριμένες ημερήσεις διατάξεις και προκαθορισμένα θέματα, να μιλάμε μεταξύ τους. Αλλά σε αυτή τη φάση ας μην ε, επικεντρωθούμε τόσο πολύ στη δημιουργία ενός επισήμου πλαισίου που θα είναι πολύ δύσκολο μετά να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιασμοί σε σχέση με, τις, με την πρωτοβουλία αυτή. Επίσης, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή. Γίνεται διπλή δουλειά με το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, με την, ε, τις διάφορες επιτροπές εκεί, ε, τον ΩΣΑ, που έχει αρχίσει επίσης μια παρακολούθηση για την χρηστή διακυβέρνηση ε, στο πλαίσιο της Επιτροπής Γκρέκο, της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, ο καθένας λοιπόν πρέπει να μπορεί να προσπαθεί να εξειδικεύεται στον τομέα του και να αποφύγουμε τις ε, αλληλοεπικαλύψεις. Και για να απαντήσω σε αυτό που είπε η κυρία ε, Φωνστόκ, οι ευρωπαϊκές αξίες είναι θεσμοθετημένες στο, στα ευρωπαϊκά κείμενα, στη, θεμελιο, στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε άλλα διεθνή κείμενα, τα οποία επιβάλλονται σε όλους και κανένας δεν μπορεί να τα θέσει ένα αμφιβόλο. Ευχαριστώ. Ο κ. Βιτάνη από την Ουγγαρία. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω την Ουγγρική θέση για το θέμα αυτό. Για μας το κράτος δικαίου είναι μια αρχή που πρέπει να προστατεύεται, αλλά για να λύσουμε την κατάσταση του κράτους δικαίου, θα πρέπει να βασιστούμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου του 2004. Θα πρέπει δηλαδή να βασιστούμε σε κοινέ αρχές. Εμείς βασιζόμαστε σε ένα διάλογο που θα χαρακτηρίζεται από τις εξή αρχές. Αντικειμενική αξιολόγηση των κρατών μελών, όχι διακρίσεις, ισότητα μεταξύ των κρατών μελών και εστίαση αμερόληπτη σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Αλλιώς τα πάντα είναι απαράδεκτα. Γίνονται απαράδεκτα. Θα πρέπει να βασιστούμε λοιπόν σε αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2004 και να αποφύγουμε τα θέματα που μας διαιρούν και προκαλούν διχογνωμίες. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου επίσης λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2016 υιοθετήθηκε ένα ψήφισμα το οποίο πρότεινε τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη δημιουργία κράτους δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτός ο μηχανισμός πάντα ενδιέφερε την Ουγγαρία και ήθελε, η Ουγγαρία θέλει δηλαδή ο μηχανισμός αυτός να έχει τα απαραίτητα μέσα για να παίξει το ρόλο του. Όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει νομική βάση. Έτσι. Άρα, τι κάνει αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα ασκεί πολιτική πίεση και ανακατεύεται, χώνεται σε εθνικές υποθέσεις. Εμείς πάντα είχαμε δείξει ανοιχτό πνεύμα. Να συζητήσουμε, να κάνουμε διάλογο. Και πάντα θα είμαστε ανοιχτοί για να κάνουμε διάλογο με σκοπό να βρούμε λύσεις. Ευχαριστώ. Έχω τέσσερις ακόμα μιλητές. Ο κ. Βόκτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω παραθέτοντας αυτά που είπατε, γιατί είπατε ότι τα αποτελέσματα των ε, συζητήσεων είναι ότι χρειαζόμαστε μηχανισμούς ε, που θα εγγυηθούν τη διατήρηση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συμφωνώ. Το ερώτημα όμως είναι ότι κατά πρώτον τι μηχανισμοί είναι αυτοί και πώς μπορούν να λειτουργήσουν αν στην Ευρώπη αυτή τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ε, ίδια για όλους, δεν ισχύουν τον ίδιο τρόπο για όλους. Ο συνάδελφος προσπάθησε να θίξει το θέμα της αποπολιτικοποίησης. Για παράδειγμα, ένας, ένας γιατρός ε, ε εγχειρίζει. Δεν έχει σημασία αν είναι αριστερός ή δεξιός ο ασθενής του. Αυτό φαίνεται όμω δεν ισχύει στην εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το κατά πόσον, για παράδειγμα, το εν λόγω άτομο είναι αριστερό ε, ή δεξιό. Εγώ στη χώρα μου, όταν ήμουν ε, πρόεδρο του NPD στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, ένας υποψήφιος αντιμετώπισε το εξής πρόβλημα. Ο παιδιατρό αρνήθηκε να φροντίσει τα δυο του παιδιά, γιατί είπε ότι ο πατέρας ε, ψήφιζε το NPD. Και είχε προτάξει το επιχείρημα ότι ε, ναι είχε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, μπορεί να είχε προβλήματα στην εφαρμογή του. Το τελευταίο μήνα στη Γερμανία είχαμε τη μεγαλύτερη, την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ε, αγωγής ε, μετά τον ε, πόλεμο 26 καταγγέλλοντες, 60 εκατομμύρια κόστος. Μετά από 3,5 χρόνια, μετά από τόσες ημέρες διαβουλεύσεων ε, διεκόπηκε η διαδικασία εξέτασης της αγωγής γιατί βγήκε στη σύνταξη ο δικαστής. Και ουσιαστικά τι έγινε, αναβλήθηκε τόσο πολύ η δικαστική αγωγή μέχρι ότου να μην είναι δυνατή η δικαστική απόφαση. Και τώρα η εισαγγελία ζητά να γίνει νέα ανάθεση των ρόλων. Τρεις χρόνια, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, υπήρχαν διαβουλεύσεις. Χάσαν τα άτομα αυτά τη δουλειά τους. Ήταν υπό εξέταση, γιατί α, μόνο και μόνο λόγω πολιτικών πεπιθήσεων στις Ουγγρικές αρχές, στις Γερμανικές αρχές, ε, υπήρξε έκδοση από τους ε, Γερμανούς τους Ούγγρους λόγω πολιτικών πεπιθήσεων μόνο και μόνο επειδή στη Γερμανία πολλοί έχουν διαφορετική άποψη. Σας παρακαλώ, λέει η όσο να ολοκληρώνετε. Ναι, κοιτάξτε. Χάνουν λοιπόν το βιό τους λόγω πολιτικών επιθύσεων Και ένα δικαστή του AFD. Και να μην μιλήσουμε καν για τους ε, στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους επειδή ήταν πατριώτες. Ε, να είναι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να μιλάμε για ισότητα. Σας ευχαριστώ κυρία Φαν Βέιζελ τώρα από τις 100 χώρες. Βέιζελ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά, αφού μπορώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας Είμαι η Άννεκε Βέζελεκ, πρόσωπος της ε, Ολλανδικής Γερουσίας. Είναι σημαντικό το ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τηρούν την ευρωπαϊκή, την εθνική νομοθεσία, αλλά και τη διεθνή νομοθεσία. Το ίδιο περιμένουμε και από τους Ευρωπαίους πολίτες άλλωστε. Η δική μου ερώτηση προς τα μέλη του πάνελ είναι γιατί δεν ξεκινάμε με έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα μεγάλο σκοπό και αυτό σκοπό αν θέλετε. Και το θέτω αυτό το ερώτημα γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι σαφές το τι ακριβώς ελέγχεται όταν μιλάμε για δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Ποιος καθορίζει το τι εννοείται ακριβώς με τους όρους αυτούς. Από ό,τι φαίνεται, αυτές οι αρχές δεν ορίζονται επαρκώς. Σας ευχαριστώ και αν θέλετε να με απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Κύριος Χάμπουλ, θα πάρει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Uh, θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις δικές μου εντυπώσεις. Τι αποκομίζω από αυτή τη συζήτηση. Πάντως αυτή η συζήτηση δείχνει σαφέστατα ότι ήταν πολύ χρήσιμος αυτός ο διάλογος Περισσότεροι, διάφοροι περιπτώσει, είπαν ότι ο διάλογος είναι καλό πράγμα, αλλά όχι η πίεση. Φυσικά υπάρχει μια έμεση πίεση, καθώς συγκρίνουμε την κατάσταση στις διάφορες χώρες. Και νομίζω ότι αυτή η έμεση πίεση είναι χρήσιμη. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Αυτός ο μηχανισμός, αν εφαρμοστεί, θα αφορά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου κυρίως. Το θέμα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλύπτεται αρκετά καλά, νομίζω, από τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι το καλύπτουμε αρκετά καλά. Σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Βεβαίω, το να μπουν στην εθνική νομοθεσία κάποια γενικά πράγματα και που προωθούν ας πούμε, κάποια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Τρίτη παρατήρηση. Το θέμα είναι εν οι αξίες μας. Ακούστηκαν πάρα πολύ. Έχουμε ένα βασικό κατάλογο πολύ ε, θεμελιακών αξιών και υπάρχει μια πιο πλήρης περιγραφή του τι εννοούμε στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βεβαίως υπάρχουν ε, ποικίλε ε, και διαφορετικές αξίες και μερικές φορές είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε πάνω σε συγκεκριμένες αξίες. Οποιοςδήποτε λοιπόν μηχανισμός όπως αυτός προτείνεται σήμερα θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στις διαδικασίες. Όχι τόσο στο περιεχόμενο των αξιών. Θα πρέπει να περιγράφει μια πορεία. Συχνά δεν θα μπορούμε να τα διαχωρίζουμε απόλυτα αυτά τα δύο, αλλά νομίζω ότι καταρχήν θα πρέπει να μιλάμε για διαδικασίες. Αυτός ο μηχανισμός να ελέγχει τις διαδικασίες. Και τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω. Ποτέ δεν υπάρχει αρκετό χρόνο το ξέρω. Το τελευταίο μου λοιπόν σχόλιο είναι το εξή. Διάφοροι από εσά είπαν ότι καλή είναι η συζήτηση, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε όλα αυτά. Όλα αυτά που αποφασίζουμε. Αυτό δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο μας θέμα. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό η εφαρμογή. Η εφαρμογή των αποφάσεων και το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς εφαρμόζεται εγείρει κάποια προβλήματα. Και το λέει αυτό κάποιος από μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα πλαίσια, ε, την έχει παραπέμψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διαδικασία επί γιατί δεν εφαρμόζει τους κανονισμούς. Δεν είναι μόνο η χώρα μου όμως, υπάρχουν και άλλες χώρες ε, οι οποίες δεν εφαρμόζουν άλλα, τμήμα, άλλα τμήματα του ευρωπαϊκού δικαίου και δεν ε, επικρέμαται αυτή τη στιγμή επάνω τους καμία διαδικασία επί παραβάκη, θα πρέπει να τις εξετάσουμε και αυτές τις χώρες, έτσι. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω στα γαλλικά με ένα γενικό σχόλιο. Το είπαν διάφοροι εσείς, η κυρία Γεβό και οι εκπρόσωποι της Γαλλικής Γερουσίας. Και τι λέει, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά με την ενιαία αγορά και θα πρέπει να ανήκει στον όγκο του, στο πλαίσιο του συνταγματικού δικαίου. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό θέμα είναι ο διάλογος και το θέμα του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το πώς θα εξασφαλίσουμε να κάποιους αποτελεσματικούς μηχανισμούς για το σεβασμό του κράτους δικαίου, έχουμε διάφορα εργαλεία. Έχουμε το νομικό κεκτημένο, έχουμε τη συνείδηση των πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τρίτον, την εφαρμογή. Για το πρώτο, το κεκτημένο μας για τη διατήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι θαυμάσιο, το είπατε. Το πρόβλημα είναι να περάσουμε από την αρχή στην πράξη, όπως είπε και ο Πορτογάλος εκπρόσωπος. Και τώρα, θα επικεντρωθώ στη συνειδητοποίηση των πολιτών. Η Ολλανδέσα συνάδελφος το εντόπισε αυτό πολύ σωστά. Φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα που έχουν οι πολίτες μας να είναι ενεργά και πρωταγωνιστικά μέλη στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με πολύ ταπεινοφροσύνη στην Κομισιόν προσπαθούμε να προωθήσουμε κάποια κατάλληλα εργαλεία. Έχουμε ετοιμάσει μια εφαρμογή που με ένα κλικ οι, ευρωπαϊκοί, οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να εξετάζουν την εφαρμογή του, των δικαιωμάτων. Επίσης, μια πλήρης πρόσβαση ε, σε κείμενα, ούτως ώστε ο πολίτης να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του. Οποιοςδήποτε πολίτης ή οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση να διαβάσει τα συγκεκριμένα δικαιώματα στο ίντερνετ είναι πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να εξασφαλίσουμε την αφύπνιση, τη συνειδητοποίηση. Αλλά είναι κάτι πολύ περίπλοκο να γίνει στην πράξη. Εύκολο να το πει, αλλά δύσκολο να το κάνει. Και σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή των δικαιωμάτων, είμαι ένα ταπεινό δημόσιο υπάλληλο. Αλλά δεν συμφωνώ με τη γνώμη, κάθε ταπεινότητα, ότι η Κομισιόν ξεπερνάει τι αρμοδιότητέ τη, ότι αναμειγνύεται σε πράγματα που δεν την αφορούν ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς ασχολείται με θέματα πολιτικής και λέει ότι η Κομισιόν δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε πολιτική συζήτηση στην Πολωνία. Τα πολιτικά θέματα στην Πολωνία είναι η δουλειά των πολιτικών της Πολωνίας και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δουλειά η δική μας είναι να διατηρήσουμε το κράτος δικαίου με βάση τις ευθύνε μας που απορρέουν από τις συνθήκες. Τελεία. Το κράτος δικαίου και το πλαίσιο για το κράτος δικαίου για μας είναι το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε την ε, υποχρέωση να μερνήσουμε γι' αυτό. Και το Μάιο, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, μια μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος με την πολωνική κυβέρνηση, ούτως ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη για να προωθηθούν οι αρχές του κράτου δικαίου. Δεν επικρίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπερβάση των αρμοδιότητων τη. Ε, την επικρίνω γιατί δεν την ε, χρησιμοποιεί στην πλήρη έκτασή του στι αρμοδιότητε αυτέ. Σα ευχαριστώ όλου πολύ. Θα κάνω κάποιε καταλεκτικέ παρατηρήσει και μετά θα σα κάνω και μία πρόταση. Δείξτε λίγη υπομονή. Πιστεύω ότι υπάρχουν βασικά κάποιε παρανοήσει για το τι πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διευκρινίσω και την τελευταία νομία εξ αυτών, ελπίζω. Το θέμα που δείξατε πολύ ημών, ποιο θα θέσει τα στάνταρτα πρότυπα, ποιο θα πει τι είναι κανονικό και τι είναι φυσιολογικό, θα μα επιβληθούν από τον εξάρτητο αυτό πάνελ εμπειροχνομόνων οποιασδήποτε αρχέ και, και πρόκειται για άτομα που δεν έχουν και δημοκρατική και πολιτική νομιμοποίηση. Όχι, όχι. Είναι σαφέστατη και κατηγορηματική η απάντηση. Όχι. Καταρχά, πολλά από αυτά τα πρότυπα ήδη υπάρχουν, έχουν ήδη οριστεί σε ευρωπαϊκέ νομοθεσίε, από την Ευρωπαϊκή Νομολογία, από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πολλά από τα πρότυπα αυτά ήδη υφίστανται και ξέρετε τι είναι αστείο, ότι όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από το δίλημα της Κοπενχάγης, ότι έχουμε δηλαδή ήδη ορίσει άρχες και πρότυπα στα κριτήρια της Κοπενχάγης. Χρησιμοποιούνται λοιπόν τα πρότυπα αυτά για να αξιολογηθεί κατά πόσο μια υποψήφια χώρα είναι έτοιμη να προσχωρήσει στην Ένωση. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε θέσει κάποια πρότυπα ήδη. Αν το θέμα είναι πώ τα εφαρμόζουμε, αυτή τη στιγμή σε μια χώρα είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Δεύτερον, Έχουμε ήδη πολλούς μηχανισμούς οι οποίοι βασίζονται σε πρότυπα όπως για παράδειγμα ο ε, πίνακας αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δικαιοσύνη. Ε, δεν πρόκειται να ε, εφεύρουμε κάτι διαφορετικό. Όσον αφορά τώρα τον περαιτέρω καθορισμό των προδιαγραφών, αυτό είναι μια κοινή διαδικασία και γι' αυτό ακριβώς πρόκειται ε, περί αυτού πρόκειται η, πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε περισσότερο να μεταγράψουμε στην πράξη αυτές τις προδιαγραφές, να είναι πιο σαφείς οι αξίες και σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Φωνστόιχ, όλοι θα συμμετέχουν στη συζήτηση, όλες οι απόψεις θα εισακούσουν ξέρω τις απόψεις σας και εσείς μπορείτε να τις εκφράσετε. Θα συμφωνήσετε ενδεχομένως μαζί μας προς αυτό. Δεν σημαίνει ότι όλα ε, είναι σχετικά. Έχουμε κάποια ζητήματα που είναι θεσμοθετημένα στις συνθήκες, όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, δεν υπάρχουν διακρίσεις για λόγους ε, φίλου, ε, αναπηρίας, ε, εθνικότητας, θρησκευτικών πεπιθήσεων κλπ. Αυτά δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Τώρα το πώς θα τα εφαρμόσουμε και τις λεπτομέρειες της μεθοδολογίας εφαρμογής είναι αυτό είναι κάτι το συζητήσιμο για το ζήτημα τώρα του πώς θα συμμετέχουν οι πολίτες. Αν διαβάσετε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει ένας πολύ διεξοδικός ε, ρόλος ε, των εκπροσώπων των πολιτών και των ε, εθνικών βουλευτών, δηλαδή και μέσω των βουλευτών αλλά και μέσω άλλων φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Έτσι προέκυψε η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε μια σειρά διαβουλεύσεων με κάθε είδους εκπροσώπων, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκκλησίες, ε, ε, κοινωνικούς εταίρους, δικαστική εξουσία, ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πάρα πολύ ευρύ, ε, ευρία ε, διαβούλευση κάναμε. Όλες οι απόψεις ακούστηκαν και έτσι φτάσαμε σε αυτή την πρόταση και αν θέλουμε να την επεξεργαστούμε περαιτέρω μαζί, αυτή είναι η ίδια προσέγγιση την οποία εγώ θα ε, υπερασπιστώ. Τελευταία παρανόηση που είναι πάρα πολύ κοινή παρεμπιπτόντος και πολύ συχνά μερικές φορές τη τις και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα κράτη-μέλη διαφωνούν. Όχι. Είναι εξαιρετικό μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συνεργάζεται περισσότερο ε, ως προς αυτό με, τα, ε, με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και το Συμβούλιο από ότι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πραγματικά είναι μία εξαίρεση. Βέβαια, έχω την πεποίθηση ότι θα υπερβούμε αυτό το σκόπελο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να βρει ένα μηχανισμό που θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να συζητήσουν λεπτομερέστερα και πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά, γιατί τώρα είναι πολύ γενική φύσεω οι συζητήσει, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ ικανοποιητικό και θα γίνει μία συζήτηση ενδεχομένως σε ένα κράτος μέλος ε, μόνο και αυτό είναι περίεργο γιατί είναι σαν να λέμε ότι αυτό το κράτος μέλος είναι αυτό το οποίο δακτυλοδεικνύουμε όλοι και κατηγορούμε ενώ υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα κράτη-μέλη. Κάτι ακόμη θα ήθελα να πω συνοψίζοντας, ε, το οποίο το ανέφερε και ο κύριος Παρασκευόπουλος. Είπε ότι χρειάζεστε, χρειαζόμαστε μία μόνιμη επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το συνδέσω με την πρόταση, με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ζητώντα από όλα τα εθνικά κοινοβούλια να ορίσουν έναν εισηγητή. Αν συνδυάσουμε αυτές τις δύο προτάσεις, εγώ θα μπορούσα να δω πώ θα μπορούσαμε να έχουμε έναν εκπρόσωπο από το Εθνικό Κοινοβούλιο κάθε κράτους μέλους, δηλαδή 28 εκπροσώπους, συν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρχει κάποιο είδου ημιμόνιμη επιτροπή, ώστε να επεξεργαστεί περισσότερο τις προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είναι πρόταση αυτό, δεν είναι νομοθεσία που εμείς άνωθεν θα τις επιβάλλουμε. Όχι, μια συζήτηση θα γίνει και θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία να προχωρήσει περαιτέρω με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Οπότε θα ήθελα να βασιστώ σε εσά, να πάτε πίσω στα Εθνικά σας Κοινοβούλια και να ορίσετε έναν εισηγητή και σε μερικούς μήνες από τώρα να ξαναβρεθούμε δεν ξέρω τώρα ποιο το είπε, ο κύριο Προντρί το είπε, δεν θυμάμαι, ότι πρέπει πιο τακτικά να συνεδριάζουμε για, ε, με, πιο συγκεκριμένε και προκαθορισμένες ημερήσιε διατάξει. Λοιπόν, θα σα αφήσω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Θα επανέλθουμε ούτω ή άλλω προ αυτό και γραπτό. Έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι τη συνεδρίασή μα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του προσκεκλημένου μα που συμμετείχαν στο πρώτο πάνελ και πάμε στο επόμενο πάνελ μας. Μισό λεπτό να βρω τα χαρτιά μου. Δεν έχω πια χαρτιά μπροστά μου. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φράνκ Έγγελ είναι σίγουρα στο δεύτερο πάνελ. Θα ήθελα να τον καλέσω να έρθει εδώ, στο Προεδρείο. Yes, so I'm inviting onto the podium. Mr. Λοιπόν, Φρανκ Έγγελ, Δίας Κράμπιτ και Μποντρί. Παρακαλώ, ελάτε εδώ δίπλα μου. Yes, please. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ε, θα ήθελα να πάρω το λόγο τώρα για να εξηγήσω ποιοι είναι οι προσκεκλημένοι μας. Ε, ο Φρανκ Έγκελ είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει τη συζήτηση, συνάδελφος του ΕΛΚ που είναι, ήταν σκιώδης εισηγητής για την ετήσια έκθεση για το ε, σύμφωνο, όπως επίσης και τώρα είναι, τίσιος, είναι εισηγητής για την ετήσια έκθεση ε, της, των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2016. Η κυρία Ντία Σαββάδη η οποία είναι από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβουλίων της Δικαστικής Εξουσίας. Ο κύριος Κράμπιτ, που είναι το δεξί χέρι του κυρίου Τίμερμανς για τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος Μπροδρή τον οποίο Ακούσαμε ε, προηγουμένω, ε, είναι από το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου. Δυστυχώ δεν έχω τα χαρτιά μπροστά μου πια και δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα για εσά. Συγγνώμη. Είναι πρόεδρος των, ε, της Επιτροπής ε, Θεσμικών και Συνταγματικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να σας καλέσω να πάρετε το λόγο με την σειρά που ανέφερα πέντε λεπτά έκαστο, κύριε Έγγελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Σοφή. Ε, είναι πολύ δύσκολο για μένα, επειδή είμαι Λοξεμβούργιος και είναι δύσκολο να διαλέξω μία λέξη, ε, μία γλώσσα για να μιλήσω, αλλά δυστυχώς η μητρική μου γλώσσα δεν είναι επίσημη γλώσσα, οπότε θα διαλέξω από τις υπάρχουσες και για την ώρα διαλέγω τα αγγλικά, αλλά δεν θα ήθελα παρακαλώ να το πάρει κανείς ως προσβολή. Θα μου ζητήθηκε να σας κάνω μια περιγραφή των θεμάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά την επόμενη έκθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν δεν με σταματήσει ένας συνάδελφος ή σκιώδης εισηγητής, θα ήθελα να είναι μία έκθεση διακυβέρνησης φέτος για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα μη κυβερνητικά ε, στοιχεία έχουν αντιμετωπιστεί και εξετάζονται συνεχώς από τόσα άλλα κείμενα ε, και ε, διατυπώσεις για ηλικιωμένους ανθρώπους, για τις μειονότητες, για τα παιδιά, για, για, για τους ανθρώπους με αναπηρίες, για, άλλους κατηγορίες, για άλλες κατηγορίες και άλλα φαινόμενα. Όμως αυτό ούτως ή άλλως όλα αυτά καλύπτονται. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα διακυβέρνησης ε, σε αυτήν την Ήπειρο και αν δεν το έχουμε ακόμη, σίγουρα θα το αποκτήσουμε. Αυτό ε, ισχύεται από δύο φαινόμενα. Πρώτον, και τα ακούσαμε σήμερα το πρωί και δεν θέλω να ε, θίξω κανέναν λέγοντάς το, αλλά η λογική της ε, των κυβερνήσεων σε, ε, σε χώρες όπως στην Ουγγαρία και, στην, και την Πολωνία δεν είναι η γενική λογική διακυβέρνησης που θα έπρεπε να ισχύει στην, Ευρω... που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε δύο κράτη-μέλη, στο μέλλον μπορούμε περισσότερα. Που ε, μπορεί ε, να προσπαθούσαν. Αν δηλαδή η Ουγγαρία και η Πολωνία ήθελαν τώρα να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα ήταν αποδεκτοί. Δεν θα μπορούσαν να προσχωρήσουν στην Ένωση με αυτά που κάνουν. Και είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να το παραγνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ότι ε, εντάξει, έχουμε φαινόμενα τα οποία πρέπει να τα αφήσουμε σε εθνικέ κυβερνήσει. Αυτέ οι εθνικέ κυβερνήσει και τα κράτη αυτά πριν από λίγο καιρό αποφάσισαν να μπουν σε μία λέσχη με συγκεκριμένου κανόνες. Και το έκαναν αυτό προαιρετικά. Δεν του υποχρέωσε κανείς. Εγώ πραγματικά ε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν μα συγκρίνουμε την Ιουγκοσλαβία, τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση δεν ρώτησε κανέναν πώ θα ήθελε να τον μεταχειριστούν. Ε, Εμεί ρωτάμε. Ρωτάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπάθησε κανεί με το ζόρι να κάνει κανέναν μέλος. Ε, όλοι ε, συγκατατέθηκαν. Έχει κάποιο σύνολο κανόνων διακυβέρνησης που αναφέρονται στη συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, και πρόκειται ε, για αξίες οι οποίες απειλούνται σε αρκετά μέρη. Δεν είναι μόνο η Πολωνία και η Ουγγαρία είναι πιο ανεπαίσθητο αυτό. Γιατί εκτός από αυτήν την απειλή που υπάρχει ως προς την ασφάλεια με την τρομοκρατία και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό, σχεδόν καθένας, καθένας από εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την τάση να κινείται προς κυβερνητικές τάσεις που θα μπορούσαν να αποβούν επικίνδυνες. Δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθώ, για παράδειγμα, σε φαινόμενα την ε, εσωτερική κατάσταση επίγουσας ε, ανάγκης ε, στη Γαλλία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μια τέτοιου είδου επίγουσα κατάσταση στην Γαλλία για να αντιμετωπίσουμε μια απειλή με την οποία θα μάθουμε να ζούμε. Ξέρω ότι και σε άλλες χώρες, όπως η δικιά μου, προσπαθήσαμε αυτή η προκήρυξη της επίγουσας ανάγκης να είναι η λύση στα προβλήματα ασφάλειας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτή όμως η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν θα μας ε, βοηθήσει εμάς, δεν θα μας ε, ε, ε, ε ούτε, ούτε, ούτε και η κανονική συνταγματική διαδικασία θα κάνει την απειλή αυτή να απομακρυνθεί. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε να κυβερνούμε με τον τρόπο με τον οποίο θα το κάναμε ούτως ή άλλως οποιαδήποτε άλλη μέρα. Αυτά είναι φαινόμενα ε, τα οποία ε, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και έχω την πεποίθηση ότι αν συνεχίσουμε να το κάνουμε και το κάνουμε βάσει αυτής της έκθεσης επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του σχετικού μηχανισμού εποπτείας, ε, πρέπει να πούμε ότι αυτό συνάδει με την ε, μόνιμη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς κάθε διακυβέρνηση που γίνεται με τον πλέον ευρωπαϊκό τρόπο. Πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας, ακόμη και σε χώρες, και το είπα στην αρχή, στις χώρες που θεωρούμε ότι οι κυβερνητικές τάσεις δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Όλοι όσοι μας λένε ότι το θεωρούν ότι αυτό είναι ε, απολύτως φυσιολογικό, έχουν κάποιο λόγο που ενδεχομένως το κάνουν και πρέπει με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να, συνε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε μεταξύ μας, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε αποφασίσει, αν υπάρχει μια ευρωπαϊκή λογική διακυβέρνηση, αν μπορούμε όλοι ακόμη να συμφωνήσουμε επί των σημείων που ε, μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Και πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να έχουμε ε, πολύ αποκλίνουσες ε, νοοτροπίες ε, για θέματα όπως ε, για παράδειγμα η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, βασικά θέματα. Αν γίνει κατάχρηση αυτής της κατάστασης για πολιτικούς λόγους, ε, μιλάμε για αμφισβήτηση που από την, αξιών που από την Γαλλική Επανάσταση έχουμε προσπαθήσει να έχουμε στην Ευρώπη η ε, δικαστική εξουσία είναι ένας από τους πυλώνες των ευρωπαϊκών κοινωνιών και βλέπουμε τώρα ότι σε πολλά μέρη υπάρχουν μια υπάρχουν τάσεις χρήσης, μια τάση χρήσης ε, δικαστικής εξουσίας για την ενίσχυση των πολιτικών σκοπών. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη και αυτή είναι και η άποψη νομίζω όλων όσων έχουν συμμετέχει, συμμετάσχει στο μηχανισμό ε, ε, ε, εποπτείας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στη διατύπωση της σχετικής έκθεσης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι κανείς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων που υποστηρίζουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τα επόμενα χρόνια λοιπόν το βασικό θα είναι μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ όλων των κυβερνήσεων διαφόρων χρωμάτων και επιπέδων για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος, μια κυβέρνηση, ένα, μια Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Και αν διαφωνούμε, μπορεί να χρειαστεί με κάποιο τρόπο να το λύσουμε αυτό. Εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, το επαναλαμβάνω και θα ολοκληρώσω με αυτό το σχόλιο, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να έχουμε δύο, τρεις, τέσσερις διαφορετικές στάσεις σε σχέση με, ε, ποια, με τη σχέση ε, της κυβέρνησης και ε, της δικαστικής εξουσίας. Αυτό δεν έχει να κάνει με την επικουρικότητα όπως πολύ συχνά λέγεται, δεν έχει να κάνει με την εθνική κυριαρχία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 50 οι διαδοχικές ε, ευρωπαϊκές κοινότητες και ενώσεις βασίστηκαν στην ε, ιδέα ότι συμφωνούμε επί ζητημάτων δημοκρατίας και λειτουργίας των χωρών μας. Αυτό είναι το μοντέλο επί του οποίου βασίστηκε, βασίστηκαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και δεν μπορούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε τόσο ε, τόσο αποκλίνουσες απόψεις, διαμετρικά αντίθετες απόψεις, ως προς αυτό. Ξέρω ότι ε, κάποιοι τον κίνδυνο κατάρρευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τον ε, συμπαθούν πάρα πολύ, γιατί δεν συμπαθούν τη λέσχη στην οποία προσχώρησαν. Όμως, αυτή δεν είναι η δική μας άποψη. Και αυτό είναι κάτι που εγώ και άλλοι σαν και εμένα το λένε σε αδιάκοπες συζητήσει που λαμβάνουν χώρα γύρω από αυτό το τομέα. Δεν μπορεί να είσαι μέσα σε μία λέσχη και όταν είσαι σε αυτή τη λέσχη να μην σέβεσαι του κανόνε και να μην κάνει τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Πρέπει κάποια στιγμή ένα κράτος μέλος να αποφασίσουν κατά πόσο διαφωνούν ή όχι με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν διαφωνείτε, πρέπει να φύγετε. Σαν το Brexit. Αυτό είναι ο τρόπο, δεν είναι αξιοπρεπέ, δεν είναι σωστό να είσαι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, να απορροφά υποστήριξη εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα ε, να επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι διάφορε απόψει που μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται. Αυτό είναι ανήθικο, πολύ απλό, πολύ απλά. Και είναι ανήθικο για τους φορολογούμενους. Αν ο φορολογούμενο το ξέρει αυτό, δεν ήταν κάτι που θα το ενέκρινε. Οπότε, συνεπώ, πρέπει να είμαστε σαφεί επί των πραγμάτων αυτών και να ξέρουμε ότι όλοι συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα σε κάποιο κράτος μέλος ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ε, κάνει τα πράγματα όπως εκείνη νομίζει σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην κυρία Δία Σαμπάντ τώρα. Ε, ακούσαμε τώρα το ερώτημα του πώς ε, ε τίθενται ε, τα, οι προδιαγραφές. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε το Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβουλίων Δικαστική Εξουσία. τι κάνει γι' αυτό, πώ συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία ε, προδιαγραφών που είναι μια συνεχή διαδικασία. Θα θέλαμε να ακούσω λοιπόν περισσότερα για τη δουλειά σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. κυρίε και κύριοι. Καταρχάς, ε, είναι μεγάλη τιμή που με προσκαλέσατε να μιλήσω σε αυτή τη Διακοινοβουλευτική Επιτροπή. Εκπροσωπώ την ENCJ, που είναι τα Εθνικά Συμβούλια για τη Δικαιοσύνη και αυτόνομα όργανα και φορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Συμβούλια για τη Δικαιοσύνη παίζουν σημαντικό ρόλο για την υπεράσπιση τη ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη ω χωριστή εξουσία από την νομοθετική και την εκτελεστική. Ε, μέσα σε διάφορα χρόνια έχει αναπτύξει το δίκτυό μα μια σειρά από πρότυπα και καλέ πρακτικέ σε διάφορου τομεί που αφορούν του δικαστέ και το δικαστικό σύστημα. Να αναφέρω ένα από αυτό το πρότυπο που είναι το ηθικό καθήκον του δικαστή να μιλάει να το, να, όταν η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, τίθενται εν κινδύνο. Δύο εβδομάδες πριν ε, είχαμε την ετήσια Γενική Συνέλευση στο Παρίσι και υιοθετήσαμε την ε, έκθεση 2016-2017 για την εξαρτησία, τη λογοδοσία και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με τον εντοπισμό δικτών ε, για μια ανεξάρτητη και λογοδοτούσα δικαιοσύνη που θα ισχύει στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών και των χωρών παρατηρητών, παρατηρητριών εντοπίζουμε και χρησιμοποιούμε τους, τους δείκτες ε, για την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα και λογοδοσία της, ε, του δικαστή, καθώς και της δικαιοσύνης εν το της και εντοπίζουμε τις προκλήσεις για να υπάρξει αυτή η ανεξαρτησία στο δικαστικό σύστημα που αντιμετωπίζουν δικαστές. Αφού χαρτογραφήσουμε ε, τα ισχυρά και τα δυνάμα σημεία, οργανώνουμε ομάδες διαλόγων όπου αναζητούμε μέσα για να διορθώσουμε τα προβλήματα. Αυτό το project ε, συγκέντρωσε τις ε, απόψεις όλων των δικαστών στην Ευρώπη για το πώς βλέπουν οι ίδιοι την ανεξαρτησία τους. Το 2000 έγινε μια έρευνα μεταξύ δικαστών ε, για δεύτερη φορά. συμμετείχαν 11.700 δικαστές από όλη την Ευρώπη και η έρευνα έδειξε ότι κατά μέσο όρο οι δικαστές θεωρούν ότι η δική τους δικαίωση η ανεξαρτησία είναι βαθμολογείται στο 8,9 στα 10 η δική τους προσωπική ανεξαρτησία έτσι, και τις χώρες τους 8,3 συνολικά. Η έρευνα αυτή αποκάλυψε έναν αριθμό άλλων σημαντικών θεμάτων, καθώς και η αντίληψη από τους δικαστές όλη την Ευρώπη ότι οι δικαστές ε, που είτε διορίζονται είτε παίρνουν προαγωγή, ας πούμε, ε, όχι όμως βάσει της ικανότητάς και της εμπειρίας τους ε, και ότι δεν είναι επαρκώς σεβαστή η ανεξαρτησία από τα άλλα θεσμικά όργανα της χώρας τους. Ε, στο πιο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο, το 447 το πρωί του 2007, για την ε, άποψη του κοινού για την εξαρτησία της δικαιοσύνης, ε, έγινε λόγος για ανάμειξη από τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις. Ήταν ο πιο συχνός λόγος για το, για το ότι υπάρχει αρνητική στάση απέναντι στη δικαιοσύνη. Να καταλάβουμε την πραγματική, τα πραγματικά όρια της δικαστικής ανεξαρτησίας είναι χρήσιμο να εξετάσουμε ε, τις ε, βασικές αρχές του, που έχει προωθήσει το δίκτυό μας. Καταρχάς, οι δικαστές θα πρέπει να διορίζονται με βάση την αξία, την αξία τους και τις ικανότητές τους. Ε, θέλω τώρα να στραφώ προς τους ε, εκπροσώπους που είναι εδώ παρόντες. Ο διορισμός των δικαστών, δικαστών είναι ένας τομέας όπου εσείς τα Εθνικά Κοινοβούλια έχετε ειδική ευθύνη. Σε πολλά συμβούλια, τμήμα των μελών του Συμβουλίου που είναι υπεύθυνοι για το διορισμό των δικαστών, οι ίδιοι διορίζονται από το Κοινοβούλιο. Το δίκτυό μας καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τον διορισμό των, μελών που δεν είναι δικαστές, ούτως ώστε να, υπάρχει να μην υπάρξει πολιτικοποίηση του, συμβουλίου, του Δικαστικού Συμβουλίου. Το δικό μου δίκτυο πιστεύει ότι αυτά τα μέλη που δεν είναι δικαστές, ε, όταν διορίζονται από το Κοινοβούλιο, η διαδικασία επιλογής, η εκλογή ή ο διορισμός θα πρέπει να βασίζεται στην αξία και να είναι διαφανής. Ε, τα άτομα αυτά τα οποία δεν είναι δικαστές θα πρέπει να έχουν υψηλό ηθικό κύρος και θα πρέπει να φέρνουν στο δικαστικό σώμα τις εμπειρίες τους, ε, τις δεξιότητές τους ε, και ούτω ώστε ε, να εξασφαλίσουμε την εκπροσώπηση και τις απόψεις των, της των πολιτών, αυτά τα μέλη που δεν είναι δικαστές δεν θα πρέπει να είναι πολιτικοί, ούτε άτομα που έχουν πολιτικές επαφές. Ε, ο δεύτερος βασικός λόγος, ε, η βασική αρχή που θα ήθελα να αναφέρω, είναι οι μεταρρυθμίσεις. Ε, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν μετά από μία του, ελάχιστη διαβούλευση με, με τα μέλη του Δικαστικού Σώματος ή το Συμβούλιο Δικαιοσύνης. Εσείς ως βουλευτές θα πρέπει να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να λογοδοτούν για αυτά τα θέματα και να συνεργάζονται με τους δικαστές και τα συμβούλια δικαιοσύνης για οποιαδήποτε δικαστική μεταρρύθμιση. Τα αποτελέσματα αυτού του project και οι εξελίξεις στην Ευρώπη δείχνει ότι είναι δύσκολες εποχές για τη δικαιοσύνη σε όλη την Ευρώπη. Ο σεβασμός ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης είναι το βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου και αυτό αμφισβητείται σε πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Το δίκτυό μου ανησυχεί ιδιαίτερω για την κατάσταση στην Πολωνία. Τον Ιανουάριο ε, του 2017 λάβαμε ένα επίσημο αίτημα συνεργασίας από το Πολωνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης, το KRS, για να το συμβουλέψουμε να μας συμβουλευτεί μάλλον για δύο νέες νομοθετικές προτάσεις. Το Συμβούλιο του Δικτύου μου ε, εκδέχει το συμπέρασμα ότι τα νομοσχέδια θα μπορούσαν να βλάψουν την, δικαιοσύνη, την εξαρτησία της δικαιοσύνης. Τον Απρίλιο το Συμβούλιο εθέτησε μια δεύτερη δήλωση επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες και λέγοντα ότι η προστασία του κράτου ε, δικαίου είναι ευθύνη και τη δικαιοσύνη, αλλά και των άλλων ε, κρατικών και επίσημων εξουσιών. Μετά από αυτή τη δήλωση, διάφορα από τα μέλη μα και του παρατηρητέ, υιοθέτησαν μεμονωμένε δικέ του δηλώσει για να εκφράσουν τις ανησυχίες για την κατάσταση τη δικαιοσύνη στην Πολωνία. Τέλο, στην ε, δήλωση του Παρισιού επαναλαμβάνουμε τι ανησυχίε μα και τονίζουμε μια βασική προπόθεση για την διατήρηση και την ενίσχυση τη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η βάση τη αμοιβαία αναγνώριση και αυτό ποιο είναι. Η ανεξαρτησία, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα κάθε ενό από τα δικαστικά ε, συστήματα και ο σεβασμό του του κράτου δικαίου. Θέλω να σα πω ότι το δικό μου δίκτυο είναι ένα από τα δικαστικά δίκτυα που αναφέρονται στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να ενισχυθεί το κράτο ε, δικαίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση καλούμεθα, κληθήκαμε μάλλον από ένα, σε μια συνάντηση το Μάρτιο από τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Τίμων μας για να εξετάσουμε την κατάσταση της πολωνικής δικαιοσύνης. Κατά την άποψή μου, η εμπλοκή του δικτύου μου στην ανάλυση της κατάστασης της δικαιοσύνης σε ένα κράτος μέλος ε, είναι πολύ σημαντική. Μία ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι προϋπόθεση να υπάρξει κράτος δικαίου. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τη σχέση μεταξύ των τριών κλάδων ε, εξουσίας. Η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία θα πρέπει να καταλαβαίνουν σαφώς τι σημαίνει δικαστική ανεξαρτησία και λογοδοσία και τι επισύρει. Το δίκτυό μου πρόσφατα καθόρισε τη στρατηγική του για την επόμενη περίοδο. Ε, ένας από τους βασικούς στόχους που θέλει να προωθήσει είναι να δώσει στήριξη για την ανεξαρτησία, τη λογοδοσία και την ποιότητα των δικαστικών συστημάτων στην Ευρώπη και να προωθήσει την κατανόηση και τον σεβασμό της δικαστικής ανεξαρτησίας. Το δίκτυό μου θέλει να το υλοποιήσει αυτό, μεταξύ άλλων στοιχείων, ξεκινώντας ένα διάλογο με τις άλλες κρατικές εξουσίες για το κράτος δικαίου και το ρόλο της δικαιοσύνης σε ένα δημοκρατικό κράτος σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δίκτυό μου θέλει να υπάρξει και μια συνέχεια στη σημερινή συνάντηση με πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίζουν ένα ουσιαστικό διάλογο για του θέματος. Στο Παρίσι, το δίκτυο υιοθέτησε μια δήλωση για την ανθεκτικότητα της δικαιοσύνης. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για ανθεκτικά δικαστικά συστήματα που θα μπορούν να αντέχουν σε εξωτερικές πιέσεις και παράλληλα να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις ξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Είναι προϋπόθεση να έχουν την κατάλληλη ε, δομή διαχείρισης και διακυβέρνησης, ε, να έχουν τα δικαστικά συμβούλια και τα συμβούλια αυτά να υποστηρίζουν οποιαδήποτε, οποιοδήποτε δικαστικό κλάδο δέχεται επίθεση και να κάνουν ό,τι μπορούν τόσο ώστε να πείσουν την ε, εκτελεστική και νομοθετική εξουσία να υποστηρίξουν δράσεις προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας. Σε ένα δημοκρατικό κράτος είναι προϋπόθεση να καταλαβαίνουμε οι μεν, τους δε, τις ευθύνες και τις, ε, ε, τα δικαιώματα των, του κάθε κλάδου κρατικής εξουσίας και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους με αποτελεσματικό τρόπο και με τρόπο που ένα σέβεται τον άλλον. Κλείνοντας, θα ήθελα να επανέλθω στο βασικό θέμα της ε, συνόδου μας. Ειλικρινά πιστεύω ότι έχουμε κοινή ευθύνη για να στηρίξουμε τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ώστε οι κοινωνίε μα να ευημερούν και να προάγουμε την ευμερία των λαών μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, παρακαλώ, κύριε Σκρεβίτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσω το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δικαιοσύνη το 2017 και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος αυτό. Το τρέχον έτος είναι ιδιαίτερο, πέμπτη έκδοση του EU Justice for All. Και γι' αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να εξετάσουμε και κάποιες τάσεις τα τελευταία χρόνια και το πώς τα συστήματα αυτά τραποποιήθηκαν από την δημοσίευση του πρώτου scoreboard του 2013. Είναι όμως και καλή ευκαιρία να αναλογιστούμε τι διδάγματα μπορούμε να εξαγάγουμε μετά από πέντε χρόνια χρήσης του εργαλείου αυτού. Και αυτή η εμπειρία θα ήταν χρήσιμη και για σας, για ενδεχόμενου νέους μηχανισμούς, για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σκοπός του scoreboard, να υπενθυμίσω, είναι κάθε χρόνο να παρέχει μια συγκριτική ανάλυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητα των εθνικών δικαστικών συστημάτων και την εξαρτησία τους. Και στόχος είναι να βελτιωθεί φυσικά η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων. Πρόκειται για μια προϋπόθεση απαραίτητη για το κράτος δικαίου για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ασκούν τα δικαιώματα τους, ενισχύονται στις δράσεις τους και μπορούν να αναπτύξουν καλές επιχειρήσεις και ένα κλίμα φιλικό προς το επιχειρήν. Γι' αυτό λοιπόν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του Ευρωπαϊκού Ετήσιου Κύκλου για την Ευρωπαϊκή στον Ευρωπαϊκό Συντονισμό των Πολιτικών και προωθείται επίση και η αξιολόγηση που γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ποια είναι τα βασικά πορίσματα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Scoreboard για το 2017 και ποιες είναι οι τάσεις που διακρίνονται. Εν συντομία η απάντηση είναι ότι υπάρχει πρόοδος τα 5 χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα και πολλές προκλήσεις. Ας δούμε τι πρόοδος έχει γίνει καταρχάς σε μια σειρά κρατών μελών που είχαμε άλλωστε κατανομάσει και στο παρελθόν. Υπάρχουν πολλές ε, προκλήσεις, υπήρχαν μόνο πολλές προκλήσεις και παρατηρούμε ότι οι δικαστικές διαδικασίες, οι δικαστικές αγωγές για εμπορικά αστικά ζητήματα έχουν καταστεί πιο Βράχυπρόθεσμες. Το 2010, για παράδειγμα, η πιο μακρά αγωγή πήρε 850 μέρες. Το 2015 η πιο μακρά αγωγή πήρε 525 ημέρες. Και σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος διαπιστώνουμε ότι η αντίληψη ε, από πλευρά των επιχειρήσεων της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος έχει βελτιωθεί ή τουλάχιστον έχει μένει σταθερή τα τελευταία πέντε χρόνια σε δύο τρίτα και πλέον των κρατών μελών. Επίσης είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η ποιότητα των δικαστικών συστημάτων εξακολουθεί να είναι υψηλή σε πιο πολλά, στα πιο πολλά κρατή-μέλη. στα μισά κρατή-μέλη παρά τις οικονομικές δυσκολίες υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευρά των πολιτών. Η έκταση του 2017 επίσης εξετάζει πιο εντελεχώς το πώς τα συστήματα αυτά είναι προσβάσιμα για τους πολίτες σε καταστάσεις φτώχειας. Για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι στα πιο πολλά κρατημέλη οι, οι πολίτες σε κατάσταση ένδυας έχουν πρόσβαση σε νομική αρρωγή σε περίπτωση που έχουν προβλήματα. Αυτή είναι γενικώ πώς η πρόοδος που έχει σημειωθεί. Τώρα, να πω και δύο λόγια για τι προκλήσεις που παραμένουν ακόμα εκκρεμείς. Το σκορμπορ του 2017 καταδείκνει ότι οι προκλήσεις έχουν να κάνουν με την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και, όπως είπε η συνάδελφος, η παρέμβαση και η πολιτική πίεση από πλευρά της πολιτικής αποτελεί το βασικό λόγο για την ε, αντίληψη ότι υπάρχει έλλειψη δικαστική ανεξαρτησία και μεροληψία. Αυτό αποτελεί σοβαρή ανησυχία και μια σειρά κρατών μελών έχουν προβεί σε δικαστικέ μεταρρυθμίσει. Αυτέ οι νέε δικαστικέ μεταρρυθμίσει θα υποστηρίξουν περαιτέρω το κρατό δικαίου και τα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, ανεξαρτησία του δικαστικού σώματο. Δεν ε, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μεταρρύθμιση ω αυτό σκοπό. Χρειαζόμαστε καλέ μεταρρυθμίσει οι οποίες πραγματικά θα ενισχύσουν την ε, ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και η αποτελεσματικότητα των δυστικών συστημάτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε μια σειρά κρατών μελών, κυρίως ό,τι αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις, τις εκκρεμείς αγωγές, backload. Σε κάποιες χώρες λοιπόν, σε 7 κράτες, ε, χώρες μέλη, υπάρχει μεγαλύτερη ο μεγαλύτερος αριθμός εκκρεμών υποθέσεων. Για πρώτη φορά φέτος το scoreboard καταδεικνύει ότι η... έχουμε σε ό,τι αφορά αγωγές για εγκληματικά, εγκληματικές ενέργειες και για ξέπλυμα χρήματος. Από, μισό χρόνο έως τρία χρόνια χρειάζεται η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Επίση η χρήση της τεχνολογίας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Χρειάζεται καλύτερη χρήση του ICT, όχι μόνο για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Να πω δύο λόγια τώρα σε ό,τι αφορά την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη αυτού του scoreboard από το 2013. Το πρώτο μάθημα που μάθαμε είναι πόσο σημαντικό είναι να γίνεται ε, αξιολόγηση στα πλαίσια της κάθε χώρας. Ε, υπάρχει μια γενική συγκριτική επισκόπηση για τα εθνικά συστήματα. Ωστόσο, η χαμηλή αποδοτικότητα βάσει των δικτών πάντα προϋποθέτει και μια καλύτερη ανάλυση, ανταλλαχέστερη ανάλυση των αιτιών. Και γι' αυτό λοιπόν γίνεται μια πιο εις βάθος αξιολόγηση ένα χώρα σε διμερή διάλογο με τις ε, εθνικές αρχές και με τους εμπλεκόμενους φορείς. Και αυτό επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίε των κρατών μελών και οι ιδιαιτερότητες του νομικού του συστήματος. Η αξιολόγηση αυτή λοιπόν παρουσιάζεται κάθε χρόνο το Φεβρουάριο στην ε, έκθεση αναχώρα η οποία δημοσιεύεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Για παράδειγμα, το 2017 σε 14 χώρες ε, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πληροφορίες για το δικαστικό σώμα στις εκθέσεις αναχώρα. Το δεύτερο πόρισμα, το δεύτερο μάθημα το οποίο διδαχθήκαμε είναι ότι δεν θα πρέπει να υποτιμούμε την πολυπλοκότητα της εξέβρεσης ε, σωστών δικτών και της συλλογής δεδομένων. Το scoreboard ε, βασίζεται σε δεδομένα που προέρχονται από μια μεγάλη ποικιλία πηγών. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι σχετικές επιτροπές, δεδομένα από τα δικαστικά δίκτυα και από τις εφιστάμενες Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Η δικαστική ανεξαρτησία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα των προκλήσεων που σχετίζονται με τα δεδομένα των 28 κρατών μελών. Πέρα από την αντίληψη της ανεξαρτησίας που προκύπτει από την έρευνα, δεν υπάρχουν ε, ακριβείς δείκτες για το πραγματικό επίπεδο της δικαστικής ανεξαρτησίας και η συλλογή των δεδομένων για την ανεξαρτησία των δικαστών από τα Υπουργεία Εσωτερικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της ε, διάκρισης των εξουσιών. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με το Συμβούλιο των ε, Δικαστικών και με τον Πρόεδρο των ε, Δικαστικών για να εισαχθεί μια διαδικασία η οποία βαθμιαία θα καθορίζει με αντικειμενικό τρόπο το πώς οργανώνονται τα δικαστικά συστήματα προκειμένου να προστατευτεί η δικαστική ανεξαρτησία σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να μεταφέρεται ένας ε, δικαστής χωρίς ε, τη συνένεση του ή της και αν ναι, υπό όρους. Αυτή η σύγκριση με τα δικαστικά δίκτυα έχει επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, πρέπει να ομολογήσουμε. Και τώρα έχουμε μία επισκόπηση των διευθυντικών εγγύσεων για τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις. Η πρόκληση η οποία παραμένει είναι να αξιολογηθεί στην πράξη η αξία της δικλείδας αυτής ασφαλείας και χαιρόμαστε όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι και το ENSG, το δίκτυο αυτό, εργάζεται επ' αυτού και ελπίζουμε ότι ε, τα μελλοντικά scoreboard θα παρουσιάσουν τα θετικά αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι στην πράξη να συλλεχθούν τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα αυτά από 28 κράτη-μέλη. Και αυτό ε, επιδεινώνονται και από πολιτικές ε, και οικονομικές σκοπιμότητες σε κάποιες περιπτώσεις. Κάποιες κυβερνήσεις δεν θέλουν να παρέχουν τα δεδομένα για θέματα νομική βάσης και για άλλους λόγους. Τέλος, το τελευταίο μάθημα το οποίο μάθαμε από την ανάπτυξη του scoreboard για τη δικαιοσύνη είναι ότι είναι σημαντικό να κινούμαστε βήμα-βήμα με την συμπερίληψη όλων των εμπλεκομένων φορέων τέτοια βαθμιαία προσέγγιση είναι ασφαλώς ακόμα πιο απαραίτητη όταν ε, έχουμε υπόψη μας την κατάρτιση ενός νέου μηχανισμού για πολύ πιο ευρύ τομεί, όπως είναι για παράδειγμα η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ελπίζω να αποβεί ωφέλιμη η εμπειρία μας και για τις δικές σας εργασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως και... Ε, εντάσσεται στη συζήτησή μας και συμβάλλει στη συζήτησή μας και μου άρεσε αυτό που είπατε με το στοιχείο του διαγωνισμού Eurovision ε, για, το, για τη δικαστική εξουσία. Ε, όπως και στη Eurovision δεν εντυπωσιάζεται πάρα πολύ ε, για... Δεν, δεν τους αρέσει πάρα πολύ ο διαγωνισμός, αλλά κανείς δεν θέλει να είναι τελευταίος. Είναι ένα διαγωνισμό στον οποίο όλοι θέλουν να τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος Μποδί έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γαλλικά. Επειδή ο κύριος Έγγελ είπε ότι δεν θα ε, χρησιμοποιήσει την ε, επίσημη γλώσσα, καμία επίσημη γλώσσα του ε, Λουξεμβούργου, ε, υπάρχει ένα ευαίσθητο θέμα στο πλαίσιο των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, όσον αφορά την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις γύρω από αυτό το θέμα πριν πω σε λεπτομέρειες και αναφερόμενος μερικές φορές στην κατάσταση της δικής μου χώρας του Λουξεμβούργου η ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ ε, σημαντική. Δεν είναι αυτός σκοπός, είναι ένα μέσο που εξυπηρετεί την αμεροληψία της εξουσίας και της ε, δικαιοσύνας. Χωρίς ανεξαρτησία δεν υπάρχει αμεροληψία των δικαστών και χωρίς την αμεροληψία των δικαστών δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η ανεξαρτησία λοιπόν δεν ε, προορίζεται ουσιαστικά προς τη δικαιοσύνη, αλλά προς τον ε, άνθρωπο που θα αναζητήσει τη δικαιοσύνη. Γι' αυτόν ε, πρόκειται, αυτόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Είναι μια δημοκρατική απέτηση, μια δημοκρατική προσδοκία και μια απαρέγκλητη πτυχή ε, του κράτους δικαίου και της διάκρισης των ε, εξουσιών. Εδώ και πάνω από τρεις ε, αιώνες, από την εποχή του Μοντεσκέ ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστές. Η διάκριση των εξουσιών σε καμία χώρα δεν είναι απόλυτη και αυστηρή όσον αφορά τουλάχιστον την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία. Ε, το γεγονός ότι υπάρχουν ε, πολιτικές πλειοψηφίες έχει σημασία, ε, έχει ως αποτέλεσμα ότι Υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία ε, μεταξύ της ε, νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας και ειδικά όσον αφορά το κυβερνητικό κομμάτι και την πολιτική πλειοψηφία σε ένα κοινοβούλιο. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η ιδανική, ιδεατή διάκριση των εξουσιών όπως τη συνέλαβε ο Μοντεσκιό. Όμως ε, η δικαστική εξουσία σε ε, αντίθεση με την νομοθετική και την ε, εκτελεστική εξουσία είναι σαφές ότι η ανεξαρτησία η λειτουργική είναι απαραίτητη σε σχέση με τις άλλες δύο και δεν μπορεί να τίθεται ένα αμφιβόλο. Αυτή η ανεξαρτησία, αυτή η πολύ μεγάλη αυτονομία της δικαιοσύνης στους διάφορους κλάδους αφορά και την εισαγγελία ε, και τους δικαστές. Ε, είναι ένα ζήτημα ευαίσθητο για πολλούς ε, ε, για πολλές χώρες, ε, δεν επιτρέπει παρέμβαση πολιτική σε, σε, σε ζητήματα δικαστικής εξουσίας ε, και συχνά αναφέρεται ως μία από τις απειλές τις πιο διαδεδομένες. Όμως εγώ πρέπει να πω ως βουλευτής ότι αυτή η απαγόρευση της παραβίασης ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης δεν ισχύει μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για την νομοθετική εξουσία. Το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν έχει ως αποστολή να ελέγχει τη δικαστική εξουσία, τη δικαιοσύνη. Πρέπει να απέχει οποιαδήποτε παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης ε, με κίνδυνο να ε, δημιουργήσει πρόβλημα στην αμεροληψία αυτής. Το αποτέλεσμα είναι ότι η δικαιοσύνη δεν έχει, σκοπό, δεν έχει σκοπό να λογοδοτήσει απευθεία στο κοινοβούλιο. Το Εθνικό Κοινοβούλιο δηλαδή δεν θα ενδιαφερόταν να συζητήσει συγκεκριμένα ε, εκρεμείς αποφάσεις ή υποθέσεις ε, με τις οποίες έχουν επιφορτιστεί οι δικαστές της χώρας του. Είναι κάτι όμως το οποίο ε, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση εξωτερική. Αυτό το δικαίωμα πρέπει οπωσδήποτε να το ε, ε, προστατεύει το Κοινοβούλιο με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, το Κοινοβούλιο πρέπει ουσιαστικά να αποκρισταλώσει στο Σύνταγμα την ανεξαρτησία αυτή της δικαιοσύνης. Σας υπενθυμίζω ότι το νέο Σύνταγμα του Λουξεμβούργου, επί το οποίο δουλεύουμε εδώ και 15 χρόνια, εν πάση περιπτώσει φτάνουμε στο τέλος τέλος του τούνελ, μέχρι το τέλος του 2018, θα αναφέρεται συγκεκριμένα όχι μόνο στην ανεξαρτησία των δικαστών, ε, αλλά ε, και την ανεξαρτησία ε, των εισαγγελέων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούν να προστατευτούν όλες οι αρχές που αφορούν τους δικαστές και την αντικατάσταση ή τη μη αντικατάστασή τους. Ε, υπάρχουν συστήματα που έχουν πολλούς δικαστές. Πρέπει να δούμε πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ ενός καλού συστήματος δικαιοσύνης και υπέρ της ανεξαρτησίας των δικαστών. Μου φαίνεται λοιπόν σημαντικό ε, το εξής ε, επειδή θα ορίζονται και από το Κοινοβούλιο σε ένα βαθμό, ε, η επιλογή πρέπει να γίνεται λαμβανομένων υπόψεων των ικανοτήτων, της ανεξαρτησίας και της ε, διαφάνειας. Ε, στις διαδικασίες λοιπόν ε, ε, του διορισμού αυτού των δικαστών υπάρχουν και ζητήματα πειθαρχικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα της λειτουργίας. Ενδεχομένως αυτό το λειτουργήμα μπορεί να το αναλάβει ένας διαμεσολαβητής που τον ορίζει το κοινοβούλιο και είναι ένας συνομιλητής ένας συνομιλητής με τη διοίκηση ε, χωρίς, βρίσκεται δηλαδή ανάμεσα στα δύο, δεν ανήκει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δεν μπορεί να παρέμβει ε, στις εκρεμείς αποφάσεις, αλλά αν διαπιστώσει ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία στη διοίκηση, στη διαχείριση της δικαιοσύνης, θα το αναφέρει στην έκθεσή του και η έκθεση αυτή βεβαίως ε, συζητείται στις ε, διάφορες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές που είναι αρμόδιες και ενδεχομένως και σε δημόσιες συνεδριάσεις αυτών των επιτροπών. Πολλές φορές μάλιστα υπάρχουν και ψηφίσματα σε σχέση με αυτό όσον αφορά την, τα προβλήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης. Τρίτον, για το, το Κοινοβούλιο το Εθνικό είναι νομοθέτης και ως νομοθέτης θα επαγρυπνά ώστε η νομοθεσία που αφορά τη δικαστική εξουσία συμμορφώνεται ε, με το Σύνταγμα, με τις διεθνείς συνθήκες και με τις ε, γενικές αρχές δικαίου. Στο Λουξεμβούργο αυτό είναι αντικείμενο ενός συνταγματικού ελέγχου ε, του Συμβουλίου Επικρατείας πριν από, το, ναι, από τον έλεγχο τον κοινοβουλευτικό ε, και υπάρχει επίση και το συνταγματικό δικαστήριο το οποίο επιλαμβάνεται του θέματο. Είναι σημαντικό αυτό να το πω ότι πολλέ φορέ οι συνταγματικοί δικαστέ είναι ε, το πρώτο οχυρό ε, ε, που έχει να αντιμετωπίσει κάποιος που θέλει να παρέμβει στη δικαιοσύνη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα πλαίσιο κράτος δικαίου γιατί διαφορετικά το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τέταρτον, το Κοινοβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό τον κρατικό, οπότε έχει μια νομοθετική αποστολή. Πρέπει το κράτος να έχει τους απαραίτητους πόρους και το προσωπικό που χρειάζεται για να μπορέσει να ασκήσει το καθήκον του. Πέμπτον, το Κοινοβούλιο ελέγχει ε, κυρίως το Κοινοβούλιο ελέγχει την κυβέρνηση. Αν, κρύβει, λοιπόν, ότι, αν κρίνει ότι η εκτελεστική εξουσία έχει παραβιάσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα ελέγχου που έχει στο μέσο, στη διάθεσή του μέσω του εσωτερικού κανονισμού του, ε, ε, Κοινοβουλίου, γραπτές αποστολές, ε, ακροάσεις υπουργών, ε, ε, σημεία ημερήσιας διάταξης που συνεδριάζει, μιας επιτροπής που συνεδριάζει δημοσίως, όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να μπορέσει να εξετάσει τα πράγματα και να μπορέσει να γνωμοδοτήσει, να ασκήσει αυτόν τον έλεγχο. Και έχουμε δει πολλές φορές ότι έχει, έχουν προσκληθεί δικαστές, είναι όμως δύσκολο αυτό γιατί οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι ε, σε σχέση με το Κοινοβούλιο, οπότε δεν μπορούμε ακριβώς να τους καλέσουμε, μπορούμε να τους προσκαλέσουμε, δεν μπορούμε να του το επιβάλλουμε, μπορούμε να του καλέσουμε, αλλά η δική τους εμφάνιση είναι μάλλον προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτική. Τους καλούμε να παραστούν λοιπόν ενώπιον του, ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου, ε, Υπάρχει πάντως αυτή τη δυνατότητα, η δυνατότητα να προσκληθεί κάποιος ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ε, φαντάζομαι ότι δεν αφορά, δεν αφορά βεβαίως εκκρεμείς υποθέσεις, απλώς ε, ε, ε, ζητήματα καθαρά πολιτικά. στο Λιξεμβούργο έχουμε τέτοιο παράδειγμα στην πρόσβαση ιστορία μας. την άνοιξη του 2013 υπήρχε μια δημόσια συζήτηση για ενδεχόμενη παρέμβαση εκτελεστικής εξουσίας μέσω ενός Υπουργού Δικαιοσύνης στη δικαιοσύνη. Άνοιξε ξανά μία έρευνα ε, για το 1980, ε, κάποια διακοδιαχείριση και είχε δημοσίως συζητηθεί το θέμα. Ε, Οπότε χρησιμοποίησαμε όλα αυτά τα μέσα που μόλις ανέφερα. Υπήρξε τελικά δημόσια συζήτηση ε, με ψηφίσματα, ε, τα οποία ψήφισαν τελικά οι εθνικοί βουλευτές Τελικά δεν έγινε βέβαια ψηφοφορία ούτε το κείμενο για την ε, παρέτηση του Υπουργού ε, ούτε το κείμενο ε, που αφορούσε την αμέλεια για την οποία επρόκειτο του, Υπουργού και ο Γενικός Εισαγγελέας παρέμεινε επίσης ο ένα δεν είναι πια υπουργό σήμερα, ο άλλο έχει συνταξιοδοτηθεί, αλλά σα δείχνω, εν πάση περιπτώσει, ότι ο διάλογο λειτουργήσε ακόμη και αν τελικά ε, δεν ήταν ε, δεν ήταν το αποτέλεσμα 100% ικανοποιητικό. Προσπάθησα να σας παρουσιάσω τα διάφορα μέσα που έχει ένα εθνικό κοινοβούλιο στη διάθεσή του για να εξασφαλίσει τη δικαιοσύνη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όμως είναι προφανές από τη μία έχουμε τα κείμενα και τα μέσα και από την άλλη υπάρχει η πολιτική βούληση του να χρησιμοποιήσει κανείς αυτά τα μέσα, αυτά τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ένα Εθνικό Κοινοβούλιο και επαφίεται τελικά στο Εθνικό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει όπως πρέπει συνετά αυτά τα μέσα. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, στους βουλευτές. Έχουμε διάφορους που ζητούν το λόγο. Η κυρία Φλωρέα από τη Ρουμανία καταρχήν. Κυρίες και κύριοι, με, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα και σε ευχαριστώ για την ευκαιρία. Είμαι αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Είναι η πρώτη μου κοινοβουλευτική θητεία και θα ήθελα να σας μιλήσω για τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Στην χώρα μου έχουμε μια υποεπιτροπή η οποία ελέγχει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε την νομοθεσία μας ή κάποια μέτρα που έχουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που πήρε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει ε, για το, για το αν γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα ή όχι. Υπάρχει και ένα άλλο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε μια ειδική επιτροπή, κοινοβουλευτική επιτροπή, που είναι μια εξεταστική κοινοβουλευτική επιτροπή. Σε αυτή την περίοδο στη Ρουμανία υπάρχει να εξελίξει μια ειδική εξεταστική επιτροπή, η οποία αναλύει την, τα αποτελέσματα των εκλογών του 2009. Εγώ συμμετέχω εκεί. Εδώ μιλήσατε για το ρόλο του Κοινοβουλίου στο διορισμό των δικαστών. Μπορώ να σας πω ότι στη Ρουμανία οι δικαστές προτείνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και διορίζονται από τον Πρόεδρο. Το Κοινοβούλιο δεν έχει κανένα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διορισμού των δικαστών. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ελέγχου του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, έναν κοινό μηχανισμό που θα δημιουργηθεί για όλα, σε όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ σας μιλάω ως πολίτης μιας χώρας που έχει υποβληθεί σε αυτόν τον έλεγχο επί 10 χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι μια οποιαδήποτε έκθεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό εργαλείο. Αν παραδείγματο χάρη η έκθεση είναι πολύ θετική, η θετική τότε η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το, ε, την έκθεση ως ε, σήμα κατατεθέντης, ας πούμε. Όμως αν είναι κακή η έκθεση αυτή, τότε η αντιπολίτευση θα επικρίνει τη δικαιοσύνη, την ε, κυβέρνηση, κατηγορώντας τη για καταχρήσεις. Επίσης, μια τελευταία παρατήρηση. Μιλήσατε για εμπειρογνώμονες. Για εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα παρακολουθούν την κατάσταση. Ποιοι θα είναι αυτοί οι εμπειρογνώμονε, ποιο θα του ε, υποδείξει διορίσει. Υπάρχει όμω και ένα άλλο πρόβλημα. Πώ ε, εξασφαλίζουν τι πληροφορίε του αυτοί οι εμπειρογνώμονε, από ποιε πηγέ. Από την εμπειρία που έχω παρατήρησα διατρέχοντας αυτές τις εκθέσεις ε, εποπτείας της Ρουμανίας από το γνωστό μηχανισμό, παρατήρησα κάποιες ασυνέπειες. Το περασμένο μήνα ο κύριος Τίμερμανς ήρθε στο Μπουκουρέστι. Εγώ ήμουνα μέλος αυτής της κοινοβουλευτικής επιτροπής που συζήτησε με τον κύριο Τίμερμανς και μην ξεχνάτε και το μηχανισμό ελέγχου της Ρουμανίας. Στη Ρουμανία συμφωνήσαμε ότι ο μηχανισμός αυτός είναι ασκηνόμενο στόχος. Δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η ιστορία στο μέλλον. Προσοχή και σύνεση. Θεωρητικά συμφωνώ με αυτό το μηχανισμό για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Θεωρητικά όμως αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και διάφορα προβληματικά σημεία ή στοιχεία. Αν ο έλεγχος και η επαλήθευση γίνεται όπως ε, έγινε στην ε, Ρουμανία, με κινητούς στόχους, με κινούμενους στόχους από χρόνο σε χρόνο, τότε δεν είμαι και τόσο πεπισμένη. Εγώ αισθάνθηκα ότι είμαστε θύμα ε, διακρίσεων με αυτή την αυξημένη εποπτεία, ας πούμε, της οποίας στόχος ήταν μόνο η Ρουμανία. Επί 10 χρόνια, αυτά τα τελευταία 10 χρόνια παρατήρησα και, το, και είδα και στον τύπο δημοσιεύματα ότι και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρόβλημα δημοκρατίας, ε, διαφθοράς και προβλήματα με το κράτος δικαίου. Και όμως δεν υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης και επιτήρησης αυτών των χωρών. Έξω και η αίσθηση ότι είμαστε θύματα διακρίσεων. Ο κ. Σιμκόμσκια από την Πολωνία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ σημαντικό. Αντίθετα από πολλές άλλες χώρες, όπου αυτός ο έλεγχος της δημοκρατίας ήταν αισθητό. Ελέγχαμε παραδείγματο χάρη τον διαχωρισμό εξουσιών ανάμεσα στο συνομοθετική και εκτελεστική εξουσία και ήταν εξαρτησία τους. Ε, στην Πολωνία μέχρι τώρα δεν είχαμε ποτέ στη διάθεσή μα ένα τέτοιο μηχανισμό παρακολούθηση και επιτήρηση. Στην Πολωνία, λοιπόν, η κατάσταση μέχρι τώρα ήταν η εξή. Είχαμε το Δικαστικό Συμβούλιο. Είναι ένα συμβούλιο που αποτελείται από δικαστέ και ο πρόεδρο αυτού του συμβουλίου διο, διοριζόταν, υποδεικνύονταν από του ίδιου του δικαστέ. Δεν είχαμε δηλαδή ε, ένα στοιχείο κοινωνικού ελέγχου ε, σε αυτό το φορέα. Οι ίδιοι δικαστέ διόριζαν τον πρόεδρό του. Χάρηκα για αυτά που είπε ο κύριος Μποντρί, που μας περιέφερσε την κατάσταση στο Λουξεμβούργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η πολωνική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης πηγαίνει ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση, με αυτή που περιέγραψε ο κύριος Μποντρί. Σε αυτή τη μεταρρύθμιση θέλουμε να δώσουμε στο Κοινοβούλιο, που είναι ο εκπρόσωπος του λαού, κάποια επιρροή στο διορισμό αυτού των, των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Έχουμε 25 δικαστές. Από τους 25, οι 15 θα επιλέγονται από το Κοινοβούλιο. Και εν συνεχεία αυτοί οι 15 δικαστές μπορούμε να πούμε ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα εκπροσωπούν περισσότερο τους α, Πολωνούς πολίτες και εν συνεχεία θα επηρεάσουν τη, για την, ε, την επιλογή των διοικητικών δικαστών και των υπολείπων δικαστών. Δεν υπήρχε αυτό πριν. Ε, προετοιμάζοντα αυτή τη μεταρρύθμιση, κάναμε μια δημόσια έρευνα. Και σε αυτή την έρευνα, το 50% των Πολωνών και πλέον εκφράστηκαν αρνητικά για την ε, λειτουργία της δικαιοσύνης στην Πολωνία. Στην έρευνα φαίνεται ότι πάνω από το 50% των Πολωνών είχαν αμφιβολία για την εξαρτησία των δικαστών. Είχαν αμφιβολία για την ε, αποτελεσματική λειτουργία του, των δικαστών και του δικαστικού συστήματος. Συχνά Α, ακούω επικρίσεις, άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Έγγελ. Ήταν πάλι επικρίσεις για τους γνωστούς υπόπτους Πολωνία και Ουγγαρία. Σας ενθαρρύνω να κάνετε αυτό που λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να επικεντρωθείτε στις δικές σας αρμοδιότητες, στα δικά σας καθήκοντα και όχι στο να κρίνετε και να επικρίνετε την κατάσταση στα κράτη-μέλη. βασιζόμενοι πού σε δημοσιεύματα του τύπου. Θα σας, ε, θα σας ε, διαφωτίσουμε πάνω σε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της μεταρρύθμισης, γιατί αφορά την δημοκρατική επαγρύπνηση της δικαιοσύνης, ούτως ώστε οι πολίτες να επηρεάζουν περισσότερο το έργο της δικαιοσύνης. Σας ε, καλώ να επαληθεύσετε αυτές τις άδικες γνώμες που εκφράζονται για τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης μας. Προτού εκφραστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Γιούρεκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Και δεν θα ήθελα να εκφραστώ για τα νομικά ζητήματα και ό,τι αναφέρθηκε σχετικά με αυτά. Αλλά αυτή η διαδικασία για την ε, εποπτεία, την παρακολούθηση της ε, του δημοκρατικού χαρακτήρα αυτό προκαλεί πάντα δυσπιστία, γιατί υπάρχουν κράτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Υπάρχουν ήδη μηχανισμοί προ την κατεύθυνση αυτή και ακριβώ αυτέ τι ε, αξίε και τι αρχές του άρθρου 2, παρακολουθούν οι μηχανισμοί αυτοί. Και το Κοινοβούλιο βέβαια μπορεί να κάνει σχετική πρόταση και το έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά να το πω αυτό προ τον κύριο Έγγελ και να κάνω και μία έκκληση αν θέλετε. Να μην υπάρξει τιμιγορία εδώ στο σημείο αυτό. Και άλλο ένα στοιχείο. Οι αρχές του άρθρου 2 πώς ε, υλοποιούνται. Πρόκειται, όπως είπε η κυρία Σπινέλη, για αξίες οι οποίες έχουν ε, επιπτώσεις σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, σχεδόν παντού. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει θέμα πολιτικού αγώνα. Για παράδειγμα, στην Κολονία υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις επιθέσεις κατά των γυναικών στην Σουηδία, στη Γερμανία και άλλες ε, περιπτώσεις που μας καταδεικνύουν πώς η αστυνομία και τα αστυνομικά όργανα δρά και πόσα ε, ενημερώνει την κοινή γνώμη. Το Πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο δεν έχει εκφράσει οποιοδήποτε σχετικό ενδιασμό. Έχουμε την 20η επέτειο της δημιουργίας ε, του Πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και αυτό πάλι αποτελεί ένα παράδειγμα του κράτους δικαίου. Πρόκειται για μια τέτοια επέτειο. Η Πολωνία πάντα αποτέλεσε στόχαστρο επιθέσεων και αιτιάσεων. Και ο αντιπρόεδρος Τίμερμαντς ο εκπρόσωπος του αντιπρόεδρου Τίμερμαντς ε, έφυγε από την αίθουσα, αλλά δεν αποτέχουμε αυτά που λέγονται για το, για το Πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο και για τη συνθήκε τη Ρώμη κτλ. Το μοναδικό κράτο στην Ευρώπη, τότε κομμουνιστικό βέβαια, που συμμετείχε στην διαδικασία αυτή. Ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς. Ε, ερωτήθηκε για τον τρόπο λειτουργίας ε, του δικαστικού σώματος. Δεν ακούσαμε όμως τίποτα σχετικό. Έγινε όμως σχετική ακρόαση για θέματα δημοκρατίας και θέματα συνταγματικά. Η Ουγγαρία και η Πολωνία δέχονται συνέχεια επιθέσεις από τις κυβερνήσεις μας σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δημοκρατικών ε, αποφάσεων για τις οποίες έχει δώσει εντολή ο λαός. υπάρχουν σοβαρέ αμφιβολίε για το κατά πόσον αυτές οι αξίες όντω αποτελούν την βάση της ε, λειτουργίας του σώματος. Και ουσιαστικά πάντα μιλάμε για μεταπρότυπα, αν θέλετε, κριτική προς τα κοινοβούλια. Και αυτά είναι και θέματα και της αντιπολίτευσης. Φυσικά μια δημοκρατία προϋποθέτει και αντιπολίτευση παλιά δεν υπήρχε πραγματική αντιπολίτευση, αλλά κάτι λοιπόν δεν λειτουργήσε σωστά. Γι' αυτό λοιπόν και απευθύνω την εκκλησία αυτή και η πρόεδρος ε, ζητά από τον ομιλητή να ολοκληρώσει. Καταληκτική παρατηρήση. Εκπροσωπώ του ε, βουλευτές οι οποίοι στο, στην εποχή του σταχισμού πολέμησαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον εκδημοκρατισμό. Αυτή ήταν η στόχη μας τότε. Και φυσικά υπάρχουν και συνάδελφοι που έχουν άλλες πεπιθήσεις. Το γνωρίζουμε αυτό. Δεν το αρνούμαστε. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, έχουμε εμπειρία και μπορούμε να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας αυτές. Και θα ήθελα να υπάρχει αλληλεγγύη και ενότητα μεταξύ βουλευτών. Ο κύριος Βιτάνη από την Ουγγαρία. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt bizottság, tekintet arra, hogy Frank Engel úr Magyarországot, hazámat érintően is. Κυρία Πρόεδρε, δεδομένου το ότι ο κύριο Έγγελε έκανε μια ρητή αναφορά για την Ουγγαρία για τη χώρα μου, θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχά, να υπογραμμίσω ότι το Κοινοβούλιο τη Ουγγαρία ω Κοινοβούλιο μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Συμβουλίου τη Ευρώπη σέβεται πλήρω την δημοκρατία και το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να γίνουν σεβαστά αυτά. Στις 17 Μαΐου το 2017 ενεκρίθη ένα ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την Ουγγαρία προκειμένου να κινητοποιηθεί το άρθρο 7 κατά της Ουγγαρίας και πρέπει να πούμε ότι αρνούμαστε όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει κανένα αποδεκτικό στοιχείο για παράβαση του κρατούς δικαίου από πλευρά της Ουγγαρίας το 2010. Και μετά, συχνές ε, είναι οι περιπτώσεις όπου ζητείται κινητοποίηση του άρθρου 7. Εμείς ε, αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι αυτό βασίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι υπάρχει ε, απειλή, ρίσκο για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση της μεταναστευτικής ε, κρίσης. Είναι διαφορετική η ζωή στην Ουγγαρία και είναι και διαφορετική νομοθετική διαδικασία. Η Ουγγαρία είναι ανοιχτή να συζητήσει όλα αυτά τα θέματα με αντικειμενικό τρόπο και να διεξαγάγει πολιτικό διάλογο αμερόληπτο για την εξέβρεση λύσεων. Και τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ουγγαρία είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε, να αναθεωρήσουμε την πολιτική της, ε, των Βρυξελών προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Yes, thank you. Just briefly to your remark that left wing... Ευχαριστώ πάρα πολύ φιλελεύθεροι και αριστεροί ε, ευρωβουλευτές ζητούν το άρθρο 7 ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως ότι συμμετείχαν και μέλη ε, του ΕΛΚ και θα ήθελα να πω, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των σοσιαλιστών ή των πρασίνων, αλλά από τη δική μου ομάδα, όταν μία κυβέρνηση, μίας ε, φιλελεύθερης κυβέρνησης ξέφευγε, επίσης την επικρίναμε. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε μία συζήτηση για ζητήματα στην τσεχική δημοκρατία, κάναμε μία συζήτηση ε, με τους Δανούς για τη μεταχείρισή τους ε, για τους, ε, προς τους ετούντες άσυλο. Δηλαδή εμείς πάντοτε προσπαθούμε να επικρίνουμε τα κακώς πεπραγμένα και δεν υπάρχει, δεν γίνεται αυτό βάσει πολιτικών πεπιθήσεων. Λοιπόν, με την αντίστροφη φορά, να, την αντίστροφη σειρά να απαντήσουμε. Πρώτα ο κύριος Μποντρή, μετά ο κύριος Κράμπιτ, μετά η κυρία Δίας και μετά ο κύριος Έγγελ θα συνοψίσει. Κύριε Μποντρή, ευχαριστώ ε, πολύ. Θα ήθελα απλώς να ε, τονίσω ότι αυτό το ε, σχέδιο του Λουξεμβούργου για το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης, το οποίο μπορεί να μην το κατάλαβε πολύ καλά ο Πολωνός συνάδελφος. Δικαστές θα συμμετέχουν. Οι δικαστές δεν ορίζονται από το Κοινοβούλιο, δεν είναι δουλειά του Κοινοβουλίου. Ε, ε, υπάρχουν δικαστές που εκλέγονται από τους ίδιους τους δικαστές, δηλαδή κάποιοι, ε, κάποιες, κάποιες, ε, κάποιοι δικηγόροι ε, θα, θα συμμετέχουν στον ορισμό των δικαστών και θα υπάρχει και ένας εκπρόσωπος των δικαστών που θα εκλεγεί από εκείνους, αλλά το Κοινοβούλιο δεν εκλέγει κανέναν. Ο κύριος Κράμπιτ νομίζω ότι είναι μια σημαντική διευκρίνηση αυτή, όπως επίσης και το γεγονός ότι όταν τα κράτη-μέλη ξεκινούν ε, μεταρρύθμιση δικαιοσύνης, ε, δεν υπάρχει παρθενογένεση, υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, μία πεπατημένη, υπάρχουν προδιαγραφές τις οποίες επεξεργάζονται τα ευρωπαϊκά δίκτυα δικαστών και είναι σημαντικό βεβαίως να υπάρχουν, ε, να γίνονται μεταρρυθμίσεις οι οποίες ε, είναι σύμφωνες με αυτές τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αναφέρομαι κυρίως στη σύσταση της Επιτροπής ε, Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2010 που θέτει, ορίζει κάποιες προδιαγραφές και έφτασαν σε αυτές τις προδιαγραφές λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των δικαστικών συστημάτων όλων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, οι δικαστές που συμμετέχουν στο δικαστικό σώμα πρέπει να εκλέγονται από τους δικαστές και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί, Γιατί βρισκόμαστε σε έναν τομέα όπου η Ευρώπη, η Μεγάλη Ευρώπη, το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης ε, σημείωσε πρόοδο σε σχέση με 40 χρόνια πριν, έχει αναπτύξει προδιαγραφές ε, οι οποίες σήμερα είναι αποδεκτές. Είναι λοιπόν σημαντικό όταν τα κράτη-μέλη ε, σκέφτονται να μεταρρυθμίσουν τα, τη δικαστική εξουσία να γίνονται σεβαστές αυτές οι προδιαγραφέ. Είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί να υπενθυμίσουμε μία ακόμη φορά ότι ένα εθνικό δικαστήριο είναι ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ένας εθνικός δικαστής είναι δικαστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτή τη στιγμή ε, εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο. Και το δίκαιο αυτό πρέπει να ε, εφαρμόζεται στο Εθνικό Δικαστήριο, γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα, και αυτό είναι θεμελιώδης δικαίωμα του καθενός, να πάει στο δικαστήριο και να ζητήσει δικαιοσύνη, η οποία διασφαλίζεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και το δικαίωμά του είναι να πάει ενώπιον ενός δικαστή που θα είναι εξάρτητος. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε οι μεταρρυθμίσεις ε, της δικαιοσύνης να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία αυτής, γιατί διαφορετικά δημιουργείται ένα πρόβλημα για την εφαρμογή του ε, δικαίου της Ένωσης. Είναι ένα κοινό πρόβλημα λοιπόν και είναι ένα πρόβλημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι ακόμη για τις κοινέ αξίες. Το άρθρο 2 αναφέρει τις κοινέ αξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια κοινή κατανόηση αυτών των αξιών που ε, απορρέουν και από την ομολογία της ε, του δικαστηρίου και του δικού μας αλλά και του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Πρόκειται για αξίες οι οποίες μπορεί να φαίνονται γενικές, όμως και πάλι Ούτε εδώ υπάρχει παρθενογένεση. Αναφέρονται αυτές ε, οι αξίες ε, στο άρθρο 2 της ε, Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ακριβώς υπήρχε μια κοινή κατανόηση του τι σημαίνουν οι αξίες αυτές. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να επενθυμίζουμε ότι αυτές οι κοινέ αξίες είναι ουσιώδου σημασία για το κοινό μα μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση είδατε ότι η διάσταση αξία είναι ένα ε, σημαντικό ε, στοιχείο ε, ένα πράγμα είναι σαφές, το μέλλον θα βασιστεί ε, στην εφαρμογή και στον τονισμό των κοινών μας ευρωπαϊκών αξιών. Το είπατε και εσείς ε, σε σχέση με τη σχετικοποίηση αυτών των αξιών. Μπορεί να έχουμε διάφορες απόψεις για την εφαρμογή τους, αλλά ξέρουμε ότι όταν υπάρχει κράτος δικαίου δεν πρέπει να υπάρχει παραβίαση της δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να τις προσέχουμε αυτές τις αξίες και να μην θεωρούμε ότι είναι απλώς κάποια γενικά μέσα που ο καθένας μπορεί να τα ερμηνεύσει κατά το δοκούν. Και εδώ υπάρχει ένα κεκτημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ντίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι το οποίο μπορεί να παρανοήθηκε ε, και το λέω για την παρέμφαση της ε, εκπροσώπου της Ρουμανίας, όταν λέω ότι τα εθνικά κοινοβούλια παίζουν σημαντικό ρόλο στον ορισμό των δικαστών, δεν εννοώ ότι ορίζουν τους δικαστές, αλλά ορίζουν τα μη δικαστικά μέλη των συμβουλίων. Εμείς καλύπτουμε τα 28 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20 από αυτά τα κράτη-μέλη, έχουν συμβούλια δικαστών ή αντίστοιχα αυτόνομα αυτό, αντίστοιχους αυτόνομους ε, φορείς. Τα άλλα οκτώ ε, επαφίεται συνήθως ε, στους, ε, στα, στους υπουργούς, στα υπουργεία και είναι παρατηρητές στο δικό μας συμβούλιο. δεν είπα ποτέ ότι τα εθνικά κοινοβούλια ορίζουν τους, τους δικαστές. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες για τις για την μεταρρύθμιση της ε, δικαστικής εξουσίας στην Πολωνία. Αλλά βάσει της πρόσφατης έρευνάς μας μεταξύ των δικαστών, εμείς ε, ζητήσαμε να απαντήσουν ανώνυμα δικαστές ε, από όλη την Ευρώπη, 12.000 δικαστές απάντησαν. Στην Πολωνία για το ερώτημα «Κατά τελευταία δύο χρόνια θεωρώ ότι η ανεξαρτησία μου ως δικαστή έχει γίνει σεβαστή από την κυβέρνηση». 74% των δικαστών που απάντησαν στην Πολωνία διαφωνούν καθέτος. Και στην ερώτηση κατά τελευταία δύο χρόνια θεωρώ ότι η ανεξαρτησία μου ως δικαστή έχει σε σεβασμού από το Κοινοβούλιο. 72% των δικαστών απάντησαν και είπαν ότι διαφωνούν. Αυτό το λέω γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα ήθελα να θέσω επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτάκι θα σας δώσω πριν ε, δώσω το λόγο στον κύριο Έγγελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ε, πάρα πολύ σύντομα. Πρέπει να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί ακριβώς μας κατηγορείτε. Στη Γερμανία οι ομοσπονδιακοί δικαστές ε, συνεργάζονται με το Υπουργείο. Στην Αυστρία το Ομοσπονδιακό Υπουργείο ορίζει τους δικαστές, στη Σουηδία επίσης επί τη βάση υποψηφιότητας ε, την οποία ε, διαχειρίζονται οι αρμόδιοι φορείς. Ε, θέλω να πω ότι αυτό, αυτή η πτυχή υπάρχει και σε άλλα συστήματα και νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό. Μήπως μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, αυτή η παρακόλληση της ανεξαρτησίας των ε, δικαστών, πού ακριβώς έγκυται. Γιατί δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι, ε, σε τι ακριβώς ε, ε, συνίσταται η, η παραβίαση της ανεξαρτησίας των δικαστών στην Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος λέει ότι δεν πρόκειται για μια συζήτηση ούτε για την Πολωνία, ούτε για την Ουγγαρία, ούτε για καμία μεμονωμένη χώρα. Απλώς υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, από ανεξάρτητους φορείς έχουν λοιπόν ακουστεί πάρα πολύ σοβαρές ανησυχίες και μεταξύ ε, αυτών βρίσκεται και η Επιτροπή της Βενετίας αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το βασικό θέμα συζήτησής μας δείχνει όμως ότι υπάρχει ανάγκη για έναν ευρύτερο μηχανισμό που θα εξετάζει όλα τα κρατημέλη ώστε να υπάρχει και σύγκριση γιατί το θέμα δεν είναι να λέμε ένα σύστημα είναι καλύτερο από το άλλο σύστημα πρέπει να έχουμε κοινέ προδιαγραφέ. Περί αυτού πρόκειται. Στι κάτω χώρε, για παράδειγμα, εμεί δεν έχουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο. Θα ήθελα να έχουμε όμω ένα συνταγματικό δικαστήριο. Παράλληλα, δεν θεωρώ ότι ο καθένα θα έλεγε ότι αυτή τη στιγμή ότι είναι μπανανία οι κάτω χώρε χωρί δημοκρατία. Οπότε διάφορα μοντέλα μπορεί να δουλέψουν. Αν δει κανεί ε, δημοκρατικά ε, μοντέλα, μπορεί να έχει ένα, ένα πλήρου εκπροσώπηση, ε, μπορεί να έχει κάποιο που δίνει περισσότερη σημασία στις εξουσίες ε, του Κοινοβουλίου ή του Προέδρου ε, της Δημοκρατίας. Ε, ε, εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχουν κάποιες κοινέ προδιαγραφές με τις οποίες όλοι θα συμμορφώνονται. Τα συστήματα μπορούν να είναι διαφορετικά. Δεν θέλουμε να πούμε ότι ένα σύστημα είναι καλύτερο από το άλλο. Κύριε Έγγελ, έχετε το λόγο για να συνοψίσετε. ως τελικό ομιλητή. Ευχαριστώ. Εντάξει. Εντάξει, όπως και ο συνάδελφος ο κύριος Μποντρή θα μιλήσω και εγώ μία από τις ε, επίσημες χώρες της ε, ε, χώρας μου. Τρεις έχουμε, οπότε τουλάχιστον μπορούμε να διαλέξουμε. Μόνο μπανανία δεν είστε εσείς στις κάτω χώρες. Ε, ενδεχομένως, ενδεχομένως ε, μια χώρα χωρίς ε, κυβέρνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να συμβεί. Άλλωστε και στο Βέλγιο ξέρουμε ότι έχει συμβεί αυτό. Τόσο καιρό δεν είχαν κυβέρνηση και συνέχισαν να λειτουργούν τα πράγματα μια χαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς κατηγορούμε την Πολωνία, την Ουγγαρία, ενδεχομένως και άλλους, ε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, κακής διακυβέρνησης που βλέπουμε σε αυτές τις συγκεκριμένες χώρες. Δεν σημαίνει ότι άλλες χώρες δεν είχαν ποτέ τέτοια προβλήματα. Ε, λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Ε, μιλάμε για παράδειγμα ε, για την ε, πολιτικοποίηση του συνταγματικού δικαστηρίου και την αποδυνάμωσή του. Θα μπορούσε βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό, αυτό καθε αυτό. Όμως η δυναμική που βρίσκεται πίσω από αυτό δεν είναι καθόλου καλή. Μπορούμε να το πούμε πολύ διαφορετικά. Να, για παράδειγμα στην Ουγγαρία η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική και το πρόβλημα τίθεται με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Έχουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την απουσία τη ευρωπαϊκής λογικής τη διακυβέρνηση. Δεν συμφωνούμε από ό,τι φαίνεται... Ε, στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε ένα θεσμικό πλαίσιο σε μία χώρα και πώς αφήνουμε τους θεσμούς να λειτουργήσουν ελεύθερα και με ανεξαρτησία. Και πιστεύουμε, και το ξέρετε γιατί σας το προσάπτουμε ε, πρώτα στην Ουγγαρία και μετά και στην Πολωνία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ξέρετε ότι εμείς εκτιμούμε ότι ε, η ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σήμαινε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε κάποια πράγματα διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν ε, τώρα ε, να αρχίσουμε να σκοτωνόμαστε ούτε να βγούνε τα μαχαίρια, όμως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές ουγγρικές, πολωνικές ή ενδεχομένως άλλων χωρών στο μέλλον που θα είναι ανεκτές ή δεν θα είναι ανεκτές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία σχεδόν ομοσπονδία στην οποία συμμετείχατε ε, με τη δική σας βούληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, μπήκε στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Η Πολωνία και η Ουγγαρία μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνώριζαν πολύ καλά τι υπήρχε μέσα. Και πρέπει να σας πω ότι θα συνεχίσουμε κατά πάσα πιθανότητα να, να έχουμε ε, ε, ε, διαμετρικά αντίθετε απόψει. Το θέμα είναι να μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι στο πλαίσιο μια Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην χρειάζεται να προσφεύγουμε σε άλλα μέσα, να μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ πραγματικά έχω ε, είμαι, είμαι ιδιασμένος με κάποιες πολιτικές. Ε, αυτή η εκστρατεία στην Ουγγαρία, να σταματήσουμε τις Βρυξέλλες. Και ε, δεν, έχω, δεν, μπορώ, δεν έχω λόγια να σας περιγράψω. Ε, και έρχονται και μου λένε τώρα ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία και ότι 1,7 εκατομμύρια ε, ερωτηθέντες απάντησαν και αυτό θα ήταν πραγματικά μια καταπληκτική επιτυχία. Μα είναι 15% του εκλογικού σώματος που συμμετείχαν. Οι υπόλοιποι εντωμεταξύ ήδη λένε στην κυβέρνησή τους... Ε, ε, ε, εμείς δεν ε, συμμετέχουμε. Και, η δημο... και το δημοψήφισμα το ίδιο πρόβλημα έχει. Εμένα κάτι μου λέει αυτό. Όταν 15% αποφασίζει και αυτό το θεωρούμε τεράστια επιτυχία, κάτι μου λέει. ο Πρωθυπουργό ο Ούγγρος είπε ότι οι Βρυξέλλες είναι υπέρ των τρομοκρατών. και αυτό αναφέρθηκε στον Ουγγρικό τύπο. Τι να σας πω, ε, δύσκολο είναι να διαβάσω τα ουγγρικά ε, και πολύ λίγος κόσμος καταλαβαίνει τα ουγγρικά, αλλά βάση περιπτώσει υπάρχουν άνθρωποι που μεταφράζουν. Πρέπει να σας πω ότι ένας πρωθυπουργό, ένας κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι η, η πρωτεύουσα, ε, η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, υποθάλπει τρομοκράτες. Συγγνώμη, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό στο πλαίσιο της υποχρέωσής της του να έχει κάποια συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτά είναι τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Εγώ είμαι υπέρ της εφαρμογής του άρθρου 7 ε, στην Ουγγαρία και σε άλλους ενδεχομένως αύριο γιατί πραγματικά υπάρχει μια διολίσθηση προς επικίνδυνα πράγματα που αν την επιτρέψουμε ε, σε 10 χρόνια ή σε 20 ή 30 χρόνια από τώρα ολόκληρη η Ήπειρος ε, θα έχει διολιστήσει προς αυτή την κακή πλευρά και θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Mm. Όχι, κλείσαμε τη συζήτηση αναγνωρίζω ότι υπάρχουν διάφορα θέματα. κάνω δύο θέματα, τα οποία ε, είναι λίγο λεπτά και προκαλούν πολλές πολεμικές ε, και συναισθηματικές εκκρίσεις. Αλλά ο Μισελ έχει απόλυτα δίκιο όταν λέει ότι αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Να συζητάμε και αυτά τα πράγματα με το συναισθηματισμό μας, αλλά με πολιτισμένο πάνω απ' όλα τρόπο και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις από κοινού. Αυτός ήταν ο σκοπός όλου αυτού του εγχειρήματο. Από να κάνουμε μια εσωτερική συζήτηση, αυτό είναι το θέμα. Γιατί αυτή η συζήτηση για την κυβέρνηση Ορμπάν γίνεται εδώ και χρόνια και έχει αρχίσει να γίνεται κουραστική για όλους, ακόμα και για την Ουγγρική κυβέρνηση. Να έχουμε αυτό το μόνιμο μπρος-πίσω, αυτό το πινκ-πονγκ ας πούμε, ναι είναι αλήθεια, δεν είναι, όχι δεν είναι αλήθεια, ναι είναι αλήθεια, όχι δεν είναι αλήθεια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αναπτύξουμε κοινά πρότυπα βάσει αυτών που υπάρχουν ήδη. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Κράβιτς, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Χτίζουμε πάνω σε κάτι. Ο κύριος Χάμπλ και ο κύριος ε, Κράβιτς είπαν το ίδιο πράγμα επί της ουσίας. Ότι η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην λειτουργία κάθε τμήματος, κάθε μέρους αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών, αλλά είναι και μια κοινότητα δικαίου. Και όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Κράβιτς, τα δικαστήρια, τα εθνικά δικαστήρια, όταν εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, γίνονται ευρωπαϊκά δικαστήρια. Επομένως θα πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε σίγουροι ότι όλοι λειτουργούν με τα ίδια πρότυπα στην ίδια βάση. Φυσικά υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Πρέπει να τις συζητήσουμε. Δεν ε, ε, πρέπει να πούμε ότι όλα είναι σημαντικά. Υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα. Και αν κάποιες κυβερνήσεις από κάποιες χώρες λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να σεβαστούμε τα πρότυπα πια, τότε ίσως θα πρέπει να χωρίσουμε το, τα τσανάκια μας. Εγώ είμαι πεπισμένη ειλικρινά ότι η πλειοψηφία των λαών και των χωρών στις οποίες αναφερθήκαμε δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Δεν θέλουν να φύγουν. Θέλουν να είναι τμήμα τη ευρωπαϊκή οικογένεια και να βρούμε λύσει μαζί. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλου να σκεφτείτε τι προτάσει που έκανα, να ιδιορίσουμε έναν εισηγητή ανά Εθνικό Κοινοβούλιο και να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση πιο μόνιμα με βάση μια ημερήσια διάταξη, όπω πρότεινε και ο κ. Μπουτρή. Πάντα να έχουμε μια ημερήσια διάταξη και έτσι να συζητάμε και να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Παίρνουμε λοιπόν την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω αφετηρία και όχι ως σημείο κατάληξης. Σας καλώ να το κάνετε αυτό. Και η τελευταία μου παρατήρηση, που είναι μια πολύ πρακτική παρατήρηση, αυτή η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί και με πιο ευχάριστο τρόπο κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει να σας αφήσω. Θα ήθελα να είμαι παρούσα και στο γεύμα, αλλά δυστυχώς ε, πρέπει να παραστώ αλλού. Και επειδή δεν μπορώ να είμαι πανταχού παρούσα ακόμα και να κλωνοποιηθώ. Πρέπει να επιλέγω. Δυστυχώς θα πρέπει να πάω τώρα ε, στην άλλη εκδήλωση, αλλά έχετε τον κύριο Έγγελ που θα, θα με εκπροσωπήσει επάξια. Και μπορείτε λοιπόν πίνοντας και τρώγοντας να τα πείτε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή συζήτηση και ελπίζω να βασιστούμε σε αυτήν και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ.